We have enough Έχουμε αρκετά μέλη πλέον στην αίθουσα. Ε, υπάρχει ένας εκπρόσωπος από κάθε πολιτική ομάδα. Καλησπέρα σας λοιπόν. Να σας παρουσιάσω τον Επίτροπο Σεύκοβιτς, ο οποίος ήταν ε, ε, πιο ακριβής από εμά και ήρθε στην ώρα του εδώ. Και πριν του δώσω το λόγο για την ομιλία του, θα ήθελα να σταθώ στο πρώτο σημείο που έχουμε στην ημερήσια διάταξη σήμερα το απόγευμα, τι ανακοινώσει τη Προέδρου σχετικά με τι αποφάσει των συντονιστών. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομη. Τα σημεία στην ημερήσια διάταξη συζητήθηκαν όλα από του συντονιστέ όσον αφορά τον ορισμό των εισηγητών για την ε, γνωμοδότηση, για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση των ωφελών ε, των περιβαλλοντικών μέτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συντάκτης της γνωμοδότησης ε, θα είναι ένα μέλος της Ευρώπης των Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών όσον αφορά τη γνωμοδότηση για τη Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το 2011. Η έκθεση ε, πηγαίνει σε κανένα συνάδελφο από τους φιλελευθέρους και για τον προπολογισμό του 2013 για το τμήμα που αφορά στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή η έκθεση ανατίθεται σε ένα μέλος ε, του ε, Ευρώπη τη Ελευθερία και Δημοκρατία. Όσον αφορά τώρα το ψήφισμα για τα δικαιώματα των ζώων, το οποίο όπω θα θυμάστε από την προηγούμενη συνεδρίαση είχαμε αποφασίσει να προτείνουμε προκειμένου να μπορέσουμε να ζητήσουμε κοινή συζήτηση στην επόμενη Σύνοδο του Στρασβούργου. Οι συντονιστές συζήτησαν το έγγραφο το οποίο εκπώνησε η Γραμματεία ε, και είναι σύμφωνοι με αυτό. Προχωρούμε λοιπόν μετά όσα συμφωνήσαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση. Είμαστε ακόμα και εν αναμονή των υποδείξεων των μελών των αντιπροσωπιών για τις αποστολές ε, που αποφασίσαμε ότι θα γίνουν ε, στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής και πιο συγκεκριμένα μέχρι το τέλος της εβδομάδος οι συντονιστές πρέπει να διαβιβάσουν στην Προεδρία τα ονόματα των μελών που θα συμμετάσχουν στην αντιπροσωπεία της αποστολής στη Γερμανία και στην Τσεχική Δημοκρατία. Ε, προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε και το θέμα που σχετίζεται στην αντιπαράθεση μεταξύ δικαιώματος στην ενημέρωση, το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε με την δημοσίευση όλων των στοιχείων ε, για τις εργασίες μας, ε, για την Επιτροπή Αναφορών ε, και το δικαίωμα στην προσωπική ζωή, το οποίο πολλές φορές επικαλούνται και οι ίδιοι πολίτες οι οποίοι απευθύνονται σε εμά. Θα υπάρχει λοιπόν ε, ε, δυνατότητα πρόσβασης μόνο για τα μέλη της Επιτροπής, τα οποία θα πρέπει από εκεί και πέρα ε, να τηρούν εμπιστευτικές πληροφορίες για τις πληροφορίες που λαμβάνουν για τους ίδιους τους πολίτες. Άρχισαμε να ακούμε και τα μέλη της άτυπης ομάδας εργασίας για την παράκτια νομοθεσία της Ισπανίας, η οποία συστήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα επίσης συναντήθηκε και με εκπροσώπους των Ισπανικών αρχών ε, η διαδικασία είναι εξελίξη, είναι θετικό το κλίμα μεταξύ των μελών της ομάδος και ε, ο διάλογος με τις Ισπανικές Αρχές και ελπίζουμε να υπάρξουν κάποιες εξελίξεις και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα το οποίο έχει αρχίσει να είναι πλέον ε, σύνηθε στην Επιτροπή μας. Η ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης θα διανυμεθεί εντός των επομένων ερών, επομένως οι συντονιστές θα εγκρίνουν την ημερήσια διάταξη εντός των επομένων νερών. Υπάρχουν όμως κάποια σημεία τα οποία αναβλήθηκαν ε, στην ημερήσια διάταξη ε, και με τα οποία συμφωνούν οι συντονιστές. Ενημέρωσα τους ε, συντονιστές και θα ήθελα να ενημερώσω και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής ότι λάβαμε και μία πρόσκληση από πλευράς ε, της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Vivian Redding, για να συμμετάσχουμε σε μια διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να ευαρθύνουμε το θέμα της ευρωπαϊκής υπηκότητας και να οργανώσουμε και μια δημόσια ακρόαση επί του ζητήματος. Βεβαίως η Επιτροπή μας δεσμεύεται να κάνει προτάσεις και ως συνήθως να συνεισφέρει ε, και σε αυτό το ε, ζήτημα, ώστε αυτή η επικοινωνία με τους πολίτες να γίνει με, το μέγιστο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ε, και να αποφέρει καρπούς. Ε, δεν υπάρχουν άλλα θέματα να σας αναφέρω από τους συντονιστές. Ολοκληρώνεται λοιπόν αυτό το σημείο και να περάσουμε στο πιο σημαντικό σημείο της σημερινής ημέρας, ε, η δήλωση του Επιτρόπου Σεύκοβιτς τον οποίο ευχαριστώ προσωπικώς και εξ ονόματος όμως της Επιτροπής μας, διότι ε, δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα θέματά μας. Μας έδωσε τη δυνατότητα να συζητήσουμε στον γύρω των ακροάσεων που κάνουν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σε όλες τις ε, επιτροπές, παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή μας δεν είναι νομοθετικού χαρακτήρα. και τα νευραλγικά σημεία για μας, κατά τη διεξαγωγή των καθηκόντων μας, υπαγορεύονται πάντα από τους πολίτες. Όπως γνωρίζει πολύ καλά ο Επίτροπος, εμείς έχουμε ε, μια μερίσα διάταξη από συγκεκριμένε προτεραιότητες, οι οποίες καθορίζονται βάσει των προτεραιοτήτων των πολιτών. Υπάρχει ανάγκη να υπάρχει συνεργασία από πλευράς ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και σε πολλές περιπτώσεις ε, σε σχέση με τα συμφέροντα των πολιτών δεν διαπιστώνουμε ότι είναι κατάλληλα προδιατεθειμένοι ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ορισμένες φορές καθυστερούν πάρα πολύ οι απαντήσεις από πλευράς τους και το περιεχόμενό τους είναι πολύ γενικόλογο. Ε, υπάρχει και ένα θέμα σε κρεμότητα το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολλέ φορέ και το έχουμε θέσει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον ίδιο τον Επίτροπο Σεύκοβιτ ε, τη ανταλλαγή ε, ε, και της επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αναφορές ή καταγγελίες που λαμβάνει απευθείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς ε, κάθε φορά που έρχεται σε επαφή ένας πολίτης μαζί μας, ε, έρχομαστε σε επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας. Δεν γίνεται όμως το ίδιο όταν ο πολίτης απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ εγώ θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο να είναι κοινέ αυτές οι αναφορές και οι καταγγελίε των πολιτών για να υπάρχουν ε, ένα πληρέστερο πλαίσιο των, ε, ε, της κατάστασης και των αναφορών που φτάνουν στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα από τους πολίτες μας. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο θα ήθελα να δείξω για τον Επίτροπο προκειμένου να μας ενημερώσει και λίγο για τις εξελίξεις είναι το θέμα της λαϊκής πρωτοβουλίας ε, πρώτο στάδιο της ε, ε, νομοθεσίας ήμασταν πρωταγωνιστές. Ξεκίνησε μια διαδικασία που έδωσε τη δυνατότητα στους, στην Επιτροπή μας να προχωρήσει αυτή την πρωτοβουλία. Ε, εμείς συμμετείχαμε ως ε, Επιτροπή Αρμόδια για τις Ακροάσεις, κάναμε μια επιλήθευση και του κανονισμού. Ε, η διαδικασία αυτή επαλήθευσης η οποία γίνεται στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων όμως ε, έχει λάβει μια διαφορετική τροπή. και ίσως η Επιτροπή μας θα αναλάβει ε, το οργανωτικό ζήτημα μαζί με τις αρμόδιες επιτροπές για το θέμα τους και αυτό φυσικά ε, μας έχει πικράνει κάποιος γιατί είχαμε θεωρήσει ότι επειδή ακριβώς δεν είμαστε νομοθετική επιτροπή θα μπορούσαμε είχα, ίσως να διαδραματίσουμε έναν αποτελεσματικό ρόλο και να μπορέσουμε να εισακούσουμε τους πολίτες ε, οι οποίοι ε, είναι ουσιαστικά εντό εισαγωγικών οι νέοι νομοθέτες ε, που προτείνουν θέματα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ένα τελευταίο σημείο το οποίο θα ήθελα να θίξω στον Επίτροπο αφορά τις αναφορές που υποβλήθηκαν σε μας για τα ευρωπαϊκά σχολεία. Εμείς έχουμε ήδη ενημερώσει τον Επίτροπο Σεύκοβιτ επί του ζητήματος. Γνωρίζει ο Επίτροπο ποια είναι τα τροτά σημεία και οι επικρίσεις από πλευρά των πολιτών ε, που ενδιαφέρονται για το ζήτημα και θα θέλαμε να ακούσουμε και μία ενημέρωση από αυτού από πλευρά Επιτρόπου για να κατανοήσουμε κατά πόσον μπορούμε να έχουμε μια λύση και αν μπορέσουμε να συνεργαστούμε ε, για να μπορέσουμε να βρούμε όλοι μαζί από κοινού τη λύση. Σα ε, δίνω λοιπόν το λόγο κύριε Σεύκοβιτ και σα ευχαριστώ για την επίσκεψή σα εδώ στην Επιτροπή μα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας και για την καλή χρονική στιγμή. Επειδή την τελευταία φορά ήμουν εδώ το Σεπτέμβριο του 2010, ε, μια εποχή όπου ακόμα βρισκόμαστε σε προπαρασκευαστικό στάδιο ε, για να οργανώσουμε τα πάντα για την ομαλή ένταξη των Ευρωπαίων πολιτών και όλα, ε, όλοι μου έλεγαν ότι όλα πρέπει να τα φροντίσουμε, πρέπει να τακτοποιήσουμε τα του οίκου μας, ότι μαζί θα πρέπει να ασκήσουμε μια φιλική πίεση στα κράτη-μέλη, και οι εσωτερικέ τους διαδικασίες πρέπει να τακτοποιηθούν, διότι όπως θα θυμάστε υπήρξαν ορισμένοι προβληματισμοί. Κατά πόσον εμείς στην Επιτροπή αλλά και τα κράτη-μέλη θα ήταν έτοιμα για την πρώτη πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών. Και δεν έχει περάσει πολύ καιρό από τότε που είχε, γίνει, είχε αρχίσει να ισχύει. Αυτή η πρωτοβουλία ήταν 1η Απριλίου, Κυριακή. Και με τα χαρά σα αναγγέλω ότι η πρώτη πρόταση για την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών έφτασε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι πολίτε χρησιμοποιήθηκαν να υποφεληθούν ε, άμεσα την πρώτη στιγμή δηλαδή για να στείλουν τις πρωτοβουλίες. Και ε, επισήμως θα ήθελα να σας αναγγείλω ότι θέλουμε αύριο, στην ε, ημέρα της Ευρώπης, ε, να καταγραφεί η πρώτη πρωτοβουλία ε, των Ευρωπαϊκών Πολιτών. Θα είναι ECI 2012-001. Επίσης είμαι πολύ ευτυχής επειδή η πρώτη πρωτοβουλία και η πρόταση για την πρωτοβουλία περιβάλλεται από μεγάλο συμβολισμό. Ονομάζεται φρατερνιτέ, δηλαδή αδελφότητα, ε, για τους νέους, για την κινητικότητα, για την Ευρώπη, πώς να χρησιμοποιηθούν αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα για καλύτερη κατανόηση των ε, διαφορετικών πολιτισμών, των εθνών, ε, προαγωγή ανταλλαγών μεταξύ των νέων, καλύτερη μόρφωση, καλύτερη εκπαίδευση για τους νέους και είμαι ευτυχής που αυτή θα είναι η πρώτη ε, πρόταση που θα καταγραφεί στα πλαίσια αυτή τη πρωτοβουλία, διότι ανταποκρίνεται στο σημερινό κλίμα και πιστεύω ότι μαζί θα στείλουμε ένα πολύ θετικό μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλά μπορεί να προσφέρει στη νέα γενιά. Είμαι ευτυχής που η νέοι, η νεολαία, που είναι η πρώτη, θα είναι η πρώτη, θα χρησιμοποιήσει αυτή την ευκαιρία, θα υποφεληθεί από την ευκαιρία και θα κάνουμε μια καλή πρόταση. Εάν δείτε τον ιστότοπο, θα δείτε ότι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα πραγματικά καταφέραμε πολλά και ευχαριστώ να ε, συνεργαστούμε με του οργανωτέ. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Θα αναγγείλω με τι προσεχείς ημέρε ε, τις αποφάσεις για τις πέντε άλλε πρωτοβουλίε ε, που θα οριστικοποιήσουν την νομική μας ανάλυση προς ενημέρωσή σας αυτή η πρωτοβουλία αφορά την κινητή επικοινωνία, τα δικαιώματα των πολιτών, την ευημερία των ζώων και την έρευνα. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα προωθηθούν χωρίς καθυστέρηση αυτές οι πρωτοβουλίες. Στην αρχή του έτους ήμουν λίγο ανήσυχος. Κατά πόσον τα κράτη-μέλη θα ήταν έτοιμα. Και όσον αφορά το ε, Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Το συζητήσαμε αυτό και πιέζει ο χρόνος, περνάει, κυλάει ο χρόνος γρήγορα. Γι' αυτό θα πρέπει να ξεκινήσουμε γρήγορα, να είναι έτοιμα τα κράτη-μέλη, να δημιουργήσουμε σωστή υποδομή στα κράτη-μέλη για ε, να προωθηθεί αυτή η πρωτοβουλία του Ευρωπαίου πολίτε. Με τα χαρά θα ήθελα να σα αναγγείλω σήμερα με την εξαίρεση της ψυχικής δημοκρατίας, όπου αναμένεται ακόμη ε, το σινιάλο του Προέδρου που θα μας επιβεβαιώσει ή θα επικυρώσει ε, δια του νόμου, όλα τα άλλα κράτη-μέλη είναι έτοιμα να ε, αναθέσουν στις αρμόδιες αρχές αυτό το έργο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας. Και ελπίζω ότι και η ψυχική δημοκρατία σε λίγες μέρες θα είναι έτοιμη να δώσει το πράσινο φως. Πρέπει να συνεργαζόμαστε πολύ στενά με την Επιτροπή σα για αυτή την πρωτοβουλία για του Ευρωπαίου πολίτε, γιατί είμαι βέβαιος ότι κυρίω οι οργανωτές που θα υποβάλουν τις προτάσεις, οι οποίες ίσως δεν θα είναι κατάλληλες για αυτή την πρωτοβουλία ε, λόγω της θεματικής τους, δηλαδή μπορεί να, να προταθούν θέματα που καλύπτονται από τη συνθήκη της Ευρατόμ. Η νομική υπηρεσία μας εξηγεί ότι πιθανόν αυτή η πρωτοβουλία θα καλύπτεται από όλα όλες τις προτάσεις σας. Αλλά είμαι βέβαιος ότι αυτοί οι οργανωτές μπορούν να στραφούν σε εσά και αν δεν παρουσιάσουν, υποβάλλουν τις προτάσεις τους στα πλαίσια της πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων πολιτών, σίγουρα είμαι βέβαιος ότι θα γίνει αυτό ε, υπό τη μορφή αναφορών. Τώρα θα με ρωτήσετε, εάν κατά πόσον δεν κάνει κατάχρηση εξουσίας η Επιτροπή για να αποφασίσει ποιες πρωτοβουλίες θα καταγραφούν, θα εγγραφούν και ποιες θα απορριφθούν. Σας υπόσχομαι ότι θα εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή όλες τις περιπτώσεις και ότι ε, θα υπάρξει ε, νομική προσφυγή εάν εν ανάγκη, εάν υπάρχει κακοδιαχείριση. Οι πολίτες μπορούν να στραφούν στο συνήγορο και ε, εσείς οπωσδήποτε κάνετε μια ένα κοινοβουλευτικό έλεγχο και συνεπώς ο Ευρωπαίος Συνήγορος θα μπορέσει να παρέμβει εν ανάγκη. Αλλά βεβαίως υπάρχει και προσφυγή, ε, δω προσφυγής. Εάν αισθάνεστε ότι η απόφασή μας δεν είναι ορθή από νομικής απόψης, μπορεί να εφεσιβάλει ε, την απόφαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ώστε να έχετε την τελευταία λέξη πάνω σε αυτό το θέμα. Όταν σας εξηγούσα τι προπαρασκευή κάναμε και πόσες προσπάθειες καταβάλαμε, προκειμένου όλα τα θέματα που έχουν σχέση με αυτή την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολίτη να παρουσιαστούν με ένα τρόπο φιλικό στο χρήστη, ε, ε, ε, βελτιώσαμε τον ιστότοπο τις ανοιχτές πηγές open source, το λογισμικό software, για τη συλλογή ε, για, της υπογραφής online και παρακολουθούμε τις τελευταίες εξελίξεις για το πώς θα χρησιμοποιήσουμε ε, τα κοινωνικά δίκτυα και υπάρχει το share button ε, στον ιστότοπο και είναι έτσι ευκολότερο να διαβιβάζονται πληροφορίες για αυτές τις πρωτοβουλίες μέσω του Twitter, του Facebook ή άλλων ε, κοινωνικών δικτύων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε οι πιθανοί οργανωτές να μπορούν να τραβήξουν την προσοχή του κοινού και να υπάρχει μεγαλύτερη διάδοση αυτού του θέματος. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή σας χειρίζεται τα κοινωνικά δίκτυα, ε, το Twitter, και τα tweets από την Επιτροπή σας είναι πολύ ενημερωτικά, πολύ χρήσιμα για μένα και νομίζω ότι πράγματι με αυτόν τον τρόπο προσελκύουμε τον ενδιαφέρον των πολιτών για αυτή την πλατφόρμα. Και με αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσουμε στο μέλλον. Κυρία Πρόεδρε, αναφέρθηκε ε, γενικά ε, στις, ε, στην εξεργασία των αναφορών το και ξέρω ότι ε, στην ετήσια έκθεσή σας για το 2011 και από ό,τι βλέπω μέχρι τώρα ε, μπορώ να πω, ε, μην το πάρετε προσωπικά, ότι η έκθεση είναι πολύ καλή και βεβαίω είμαι ευτυχή που αναφέρεται η εξαιρετική συνεργασία μεταξύ τη Επιτροπής και της δικής σας, τη Κομισιόν τη Επιτροπή σα, και παρακολούθησα με προσοχή αυτά που είπε η κυρία Πρόεδρο. Πράγματι υπάρχουν τομεί όπου μπορούμε να βελτιωθούμε πρέπει να προχωράμε πιο γρήγορα, αλλά μερικές φορές υπάρχουν νομικοί περιορισμοί, πίεση, άλλες φορές υπάρχει ε, φόρτος εργασίας. Σας ε, διαβεβαιώνω όμως ότι θα έχουμε την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση στις αναφορές σας και στα αιτήματα της Επιτροπής σας και θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ένα θέμα ε, στο σχέδιο του κ. Τσίτσεστερ που αφορά ε, την ημέρα εκείνη, ε, ε, τις εξελίξεις. Δηλαδή το σχέδιό σας να βελτιώσετε τις απευθείας επαφές με ε, τους πολίτες, τη διασύνδεση με τους πολίτες. Και γι' αυτό αναφέρθηκα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ένας νέος τρόπος για να προχωρήσουμε διότι υπάρχουν 500.000 πιθανοί πελάτες και η ικανότητα να διεκπαιρεώνεται χιλιάδες αναφορές το χρόνο, αυτό απαιτεί ε, ε, μια καλή διασύνδεση. Αυτό το αισθανόμαστε παντού και υπάρχει αυτή η ανάγκη σε όλα τα επίπεδα της ευρωπαϊκής διοίκησης. Πρέπει να δούμε τι καινούρια μέσα υπάρχουν, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τη νέα τεχνολογία και με πιο αποτελεσματικό τρόπο. μέσα στο σύστημα εσωτερικής αγοράς ε, έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα ε, ελπίζουμε να γίνει αποτελεσματικότερο στο μέλλον και εκτιμώ το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναζητά ε, πιο σύγχρονα μέσα για τη βελτίωση της επικοινωνίας με τους πολίτες. Εάν μου το επιτρέπετε κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ολοκληρώσω με μία πληροφόρηση το Ευρωπαϊκό Σχολείο και σας είμαι πραγματικά υποχρεωμένος επειδή θίξατε αυτό το θέμα σήμερα. Εδώ χρειαζόμαστε πράγματι την βοήθειά σας. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συνέχεια παρουσιάζεται ε, στο γραφείο μου, διότι ε, περνάμε δύσκολες στιγμές ε, στη γενική διακυβέρνηση και στην διαχείριση των ευρωπαϊκών σχολείων. Παρακολουθούμε από κοντά τον τρόπο με τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο ε, υιοθετούσε τις αποφάσεις στην αρχή του χρόνου και επίσης υποστηρίξαμε την πρόταση προπολογισμού για το 2013 που για τα σχολεία τύπου 1 και τύπου 2, 2 ε, ε, έχει μια αύξηση 8%. Υπήρξε σκεπτικισμός μεταξύ των κρατών μελών κατά πόσον αυτή η αύξηση δικαιολογείται, μήπως είναι πολύ μεγάλη αύξηση το 8%. Γι' αυτό και στρέφομαι, ε, ζητώ στις υπηρεσίες, ε, ε, τις, ζήτησα στις υπηρεσίες Γενικής Διεύθυνσης Πόρων και Προπολογισμού να εξετάσουν όλες τις γραμμές του προπολογισμού. Και θα ήθελα να σας πω ότι η Επιτροπή υποστηρίζει το σχέδιο προπολογισμού όπως προτάθηκε, διότι χρειάστηκαν πολλές μεταρρυθμίσεις πέρσι. Κάναμε ελέγχους αποτελεσματικότητας στα ευρωπαϊκά, στα ευρωπαϊκά σχολεία και νομίζω ότι οι διευθυντές των ευρωπαϊκών σχολείων ε, κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες. Συγχρόνως όμως πρέπει να δούμε και την πραγματικότητα. Έχουμε περισσότερα παιδιά στα σχολεία υπάρχουν αυξανόμενα προβλήματα με ε, τους βοηθούς ε, των καθηγητών. Uh, uh, Τις αποσπάσεις των καθηγητών. Και το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να αναζητούμε μερικές φορές καθηγητές στην τοπική αγορά, πράγμα το οποίο κοστίζει πολύ και δεν έχει ε, δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη στον προπολογισμό. Συγχρόνως γνωρίζετε ότι φέτος θα έχουμε ένα σχολείο στο Λάκεν, ένα στο Λουξεμβούργο. Και σήμερα μάθαμε ότι δεν αρκούν, διότι τα ευρωπαϊκά σχολεία έχουν υπερπληθυσμό, έχουν πάρα πολλά παιδιά. Λοιπόν, η δημιουργία πέμπτου σχολείου στην, στις Βρυξέλλες είναι ένα μόνιμο σημείο στην ημερήσια διάταξη και προσπαθούμε να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις με τις βελγικές αρχές. Το αίτημά μου λοιπόν προς εσάς είναι να στηρίξετε την πρόταση του προπολογισμού όταν ε, πλέον ε, σταλεί στη Δημοσιονομική Αρχή για να εξηγηθεί στα κράτη-μέλη και σε εκπαιδευτικές αρχές εκεί ότι τα ευρωπαϊκά σχολεία είναι ένας πολύ σημαντικός σύνδεσμος ώστε τα παιδιά και οι θύνοντες να δια... Να δια... τα, εκπαιδευτικά στελέχη να διατηρήσουν την επαφή με την κουλτούρα τους, με τη γλώσσα του, με την ιστορία της χώρας και δεν υπάρχει υποκατάστατο άλλο από τα ευρωπαϊκά σχολεία στο ευρωπαϊκό σύστημα. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα σε λίγες εβδομάδες, διότι λόγω της κατάστασης έγραψα σε όλα τα Υπουργεία Παιδείας και μάλιστα πήγα στο Συμβούλιο της Εκπαίδευσης και εξακολουθώ να στέλνω ερωτηματολόγια σε όλους τους μόνιμους αντιπροσώπους της Βρυξέλλες με συγκεκριμένα ερωτήματα, δηλαδή πώς θα θέλαν να αλλάξει η κατάσταση. Τώρα λαμβάνουμε τις απαντήσεις και θα πρέπει να καταλήξουμε σε ορισμένα συμπεράσματα για το μέλλον. Και αν ενδιαφέρεται η Επιτροπή σας για αυτό το θέμα, με τα χαρά να σας δώσω πιο λεπτομερείς πληροφορίες. Διότι νομίζω ότι είναι φανερό ότι με τα προβλήματα ε, που προκύπτουν με τις αποσπάσεις των καθηγητών θα έχουμε δύσκολες καταστάσεις ε, σε δύο-τρία χρόνια. Δεν πρέπει να περιμένουμε ε, να φτάσει αυτή η στιγμή, αλλά πρέπει να βρούμε από τώρα λύσεις. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε, που περιλάβετε αυτά τα τρία σημεία στην ημερήσια διάταξη και ευχαριστώ πολύ που είχατε την καλοσύνη να με ακούσετε για, ένα τόσο, για μια τόσο μεγάλη εισαγωγή. Τώρα είμαι έτοιμο για τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο Σεύκοβιτς να ξεκινήσουμε με τους συναδέλφους για ερωτήσεις. Η κυρία Άουκεν καταρχήν. Ε, Ευχαριστώ πολύ για την πολύ θετική στάση σας στην Επιτροπή και ειδικότερα εφόσον είστε ο ε, Επίτροπος για τη σχέση με τους πολίτες και εμείς ε, όντας η Επιτροπή των Πολιτών, ε, είναι μεγάλη χαρά μας που βρίσκεστε εδώ. Όσον αφορά την όλη επικοινωνία μεταξύ των πολιτών και εμών, της Κομισιόν του Κοινοβουλίου κτλ. Ε, να σας πω καταρχάς ότι έχουμε την έκθεση της Γιουρή για την καλή ε, διοίκηση και έχουμε εδώ τον ε, εισηγητή της νομοδότησης. Ελπίζουμε να δώσετε κάποια στοιχεία ε, για τις διαδικασίες, γιατί χρειαζόμαστε καλές και συγκεκριμένες παγιωμένες διαδικασίες μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των πολιτών. Παρακαλώ ζητήστε από το Προεδρείο να κλείσουν το μικρόφωνο, γιατί κάνει παρεμβολές. Ελπίζω να λάβετε υπόψη σας ε, και την αρχή των υπηρεσιών, ε, δηλαδή το να επικεντρωνόμαστε στις ανάγκες των πολιτών είναι προς όφελος όλων μας, όλης της διοίκησης. Κάνουμε κάποια πράγματα λοιπόν όχι για να προστατεύσουμε τη διοίκηση, αλλά για να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες. Δεύτερον, ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά στην οδηγία για την ε, μελέτη ε, αξιολόγηση περιβαλλοντικών κινδύνων. Υπάρχει λοιπόν ε, αυτή η πρόκληση και πραγματικά δεν μπορούμε να αντιδρούμε σε όλες τις καταστροφές που λαμβάνουν χώρα. Ε, τότε είναι πολύ αργά. Θα είναι καλό λοιπόν να μπορούμε να δρούμε πριν είναι πολύ αργά. Το δεύτερο ερώτημα Naughty ε, είναι η πρόσβαση στα έγγραφα που μας ενδιαφέρει πολύ. Ε, στο Κοινοβούλιο έχουμε αναφέρει επανειλημμένως ότι θέλουμε να δούμε τι γίνεται με τη βελτιωμένη ε, νομική βάση στις παλιές ε, συνθήκες και τι γίνεται με την πρόσβαση στα έγγραφα. Θα πρέπει λοιπόν να ρισκάρουμε να να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί αλλιώς θα μπορούμε να ρισκάρουμε την χειροτέρευση, την επιδείνωση του 1049. Έχετε λοιπόν ε, την ισχύ να το κάνετε και σας παρακαλώ να ακούσετε τα αιτήματα των πολιτών. Όσον αφορά στις διαδικασίες επί παραβάση, ελπίζω πάρα πολύ η Κομισιόν να έχει ξεκινήσει πλέον να βάζει στην ιστοσελίδα της πότε τελειώνει μία διαδικασία έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορεί ο καθένα να μπει, να δει τι συνέβη, ποιε ήταν οι ερωτήσεις που απαντήθηκαν κτλ. Έτσι λοιπόν ε, θα είναι στα σίγουρα στην ιστοσελίδα μετά τη διαδικασία, αλλά θα πρέπει να τονίσετε και στα κράτη-μέλη ότι εξαρτάται από τα κράτη-μέλη αν θέλουν να αναρτούν αυτά τα στοιχεία εκ των προτέρων. Γιατί έτσι θα κάνουν καλή εντύπωση στους πολίτες. Ε, ε, εσείς αποφασίζετε ε, ε, είναι ο νόμος που αποφασίζει ότι μπορείς ή δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Ο νόμος όμως είναι ξεκάθαρος και ως προς το ότι εάν το κράτος μέλος θέλει να υπάρχει άμεση πρόσβαση, αν υπάρχει περίπτωση δηλαδή ε, εκπλήρωση υποχρεώσεων στην παλιά συνθήκη, τότε να μπορούν να ε, το κάνουν. Από αυτού εξαρτάται λοιπόν, από τα κράτη-μέλη. Θα ήταν καλό λοιπόν να το τόνιζε αυτό η Κομισιόν στα κράτη-μέλη. Να μην τους δίνετε την εντύπωση ότι είναι άτακτα παιδιά και υπερβολικοί όταν το κάνουν αυτό. Θα σας ε, ε, ευχαριστούσαμε πολύ ε, γιατί έτσι θα είχαμε μια αξιόπιστη επικοινωνία με τους πολίτες. Ευχαριστούμε ο Πίτερ Ιάρ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και ευχαριστώ που στην ουσία έχετε επαναλάβει τη θετική σας στάση σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Ε, συνεχίζουμε τον ε, διάλογο, ε, όντας ε, υπεύθυνοι για τα ίδια θέματα, δηλαδή τις, τα παράπονα που, των πολιτών που θέλουμε να τα τακτοποιήσουμε και θα είναι καλό πάντοτε, και είναι καλό πάντοτε εάν ε, στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, λύνονται τέτοια θέματα γιατί αυτό δεν είναι μόνο μια ζωντανή δημοκρατία αλλά και μια ζωντανή Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, έχω κάποιες ερωτήσεις. Ε, το θέμα των ευρωπαϊκών σχολείων, τα είπατε κι εσείς. Έχετε την πλήρη υποστήριξη από την Επιτροπή μας. Έχει ήδη η Επιτροπή μας ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Υπήρξαν και κάποιες αναφορές σχετικά. Κάτι που με, ας πούμε, ενοχλεί ε, σε αυτή την ιστορία προσωπικά είναι το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη Ε, δεν έχουν τόσο πολύ συνειδητοποιήσει ότι το Ευρωπαϊκό Σχολείο είναι το δικό τους παιδί. Ε, χρειάζεται λοιπόν ε, η, η, η, η χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, αλλά πρέπει να δώσουν και κράτη-μέλη κάτι. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε αυτή την συμμετοχή τους και θα ήθελα πραγματικά να αναγνωρίζουν λίγο περισσότερα τα κράτη-μέλη το ρόλο των ευρωπαϊκών σχολείων γιατί αυτούς, σε αυτά ανήκουν στην ουσία τα ευρωπαϊκά σχολεία. Το επόμενο θέμα, η μέθοδοι εργασίας της ε, Επιτροπής Αναφοράς κατά την ε, επεξεργασία των αναφορών. Έχουμε, ας πούμε, τον πολίτη, ο οποίος καταθέτει μία, ένα παράπονο, μία αναφορά, μια καταγγελία. Έρχεται αυτή στην Επιτροπή καταρχάς ε, υπάρχει πληροφόρηση και μετά συζητούμε το θέμα στην Επιτροπή. Ως εδώ καλά. Αυτό που θα ήθελα θα ήταν ε, στο ενδιάμεσο να υπάρχει ένας διάλογος, γιατί πολύ συχνά ε, λέμε ε, ως επικεφαλίδα ότι όσο το γρηγορότερο τόσο καλύτερα, όμως Πολλές φορές οι πληροφορίες μας ε, δεν είναι ενημερωμένες λόγω αυτού. Θα έπρεπε ε, Λοιπόν, καλύτερα αντί να έχουμε έναν αντιπρόσωπο εδώ της Κομισιόν στη συζήτησή μας ε, στην Επιτροπή, να υπάρχει ε, ούτως ή άλλως πριν ένας διάλογος, πριν έρθουν οι απαντήσεις στην Επιτροπή. Οπότε να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις ε, αν κάτι μας λείπει λοιπά Επίσης ιδιαίτερα σημαντικό είναι και λυπάμαι που πολλές φορές λέω μερικές φορές αλλά τέλος πάντων είναι αρκετά συχνά ε, να συζητάμε ένα θέμα εδώ στην Επιτροπή Αναφοράς έρχεται προσωπικά ο αναφέρον και δεν είναι ιδιαίτερα ωραίο όταν γίνεται η συζήτηση εδώ ενώπιον του ε, καλό είναι να το είχαμε ήδη συζητήσει. Θα ήταν λοιπόν μια καλή ιδέα αν υπήρχε αυτή η καλή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής μας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να μην επαναλάβω αυτά που είπε ο συνάδελφος. Ε, για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, όπως και εσύ. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα πράγματα, όλες οι πρωτοβουλίες που σχετίζονται με αυτό καταλήγουν εδώ στην Επιτροπή Αναφορών όταν υπάρχουν παρελήψεις και νομίζω ότι ε, το θέμα αυτής, της, αυτών των πρωτοβουλειών των πολιτών είναι κάτι που θα απαιτούσε περισσότερη δουλειά να γίνει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Η κυρία Κίνγκα Γκόντς, ευχαριστώ. Ένα σχόλιο και δύο ερωτήσεις. Καταρχάς σας ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας και για την, τα όσα μας αναφέρετε. Με χαρά άκουσα ότι η πρώτη ευρωπαϊκή ε, πρωτοβουλία πολιτών, η οποία θα ξεκινήσει, είναι και συμβολικού χαρακτήρα, ε, διότι θα ε, αφορά τις συνδέσεις και ούτω καθεξής. Και επίσης θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε με τις πρωτοβουλίες εδώ στην Επιτροπή που δεν ε, ε, πληρούν τις ε, προϋποθέσεις μιας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, διότι είμαι βέβαιη ότι θα δημιουργήσουν πολύ σημαντικά ερωτηματικά και γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει καλή συνεργασία στο μέλλον μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επιτροπής Αναφορών, ώστε κατά κάποιον τρόπο να δοθεί μια επαρκώς θετική απάντηση σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες δεν συγκεντρώνουν αρκετές υπογραφών, αλλά είναι αρκετός ο αριθμός των υπογραφών και ικανός ώστε να απαιτείται μια κατάλληλη απάντηση, ε, ίσως όχι από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά που θα ασχολείται με τα σημαντικά ζητήματα. Αναφερθήκατε και στα ευρωπαϊκά σχολεία μία από τις ε, ε, συνήθεις επικρίσεις είναι ότι τα παιδιά με ειδικέ ανάγκες δεν μπορούν να γίνουν δεκτά στα εν λόγω σχολεία διότι δεν υπάρχουν επαρκείς ε, ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι. παρά το γεγονός ότι είναι σαφής ε, η προσδοκία ότι αυτοί που εργάζονται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και έχουν άτομα με συγκεκριμένες ε, ανάγκες θα πρέπει να μπορούν να προσφέρουν και την κατάλληλη παιδεία στα παιδιά τους. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν και την άποψή σας για το κατά πόσον αυτή η αύξηση στον προπολογισμό επαρκεί για να αντιμετωπίσουμε και αυτό το πρόβλημα, το οποίο επανέρχεται συνεχώς. Το επόμενο ερώτημά μου είναι ένα ερώτημα που έλαβα από τον Μάικολ Κάσμαν, ο οποίος δεν μπορεί να παραστεί σήμερα και μου ζήτησε να θέσω το ερώτημα αλλά ε, το ανέφεραν και οι προλαλήσαντες, αφορά το θέμα της διαφάνειας. Κατά πόσον ε, ε, θεωρείτε εσείς, διότι ο Μάικολ Κάσμαν είναι ο εισηγητής για την αναθεώρηση του κανονισμού για την δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα και εξ όσων γνωρίζω από την επιστολή του, Τώρα ξεκινάει ο τριμερής διάλογος με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επειδή εσείς είστε ο αρμόδιος ε, για τις ε, διοργανικές σχέσεις, θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας την άποψη για το πώς ε, βλέπετε την κατάσταση στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κατά πόσον μπορεί να βελτιωθεί η διαφάνεια. Ε, ήταν δική του μεν η ερώτηση, αλλά θα ήθελα να ακούσω και εγώ την άποψή σας από αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Χέφνερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, διότι ο συντονιστής μας ήδη ανέφερε τρία σημαντικά θέματα. Θέλω πολύ απλά να μιλήσω σύντομα για την ε, ε, πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών και εσά, κύριε Σευκοβίτς να σας ευχαριστήσω ε, να ευχαριστήσω το επιτελείο σας για την υποστήριξη που μας δώσατε με την εργασία σας σε αυτό. Βλέπετε τώρα ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες χρησιμοποιούν αυτό το νέο δικαίωμα και εμείς, ε, από εμάς εξαρτάται τι θα προκύψει από αυτό. Εμείς ε, στο Κοινοβούλιο αλλά και εσείς στην Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις δικές μας δυνατότητες για να δείξουμε στους πολίτες ότι παίρνουμε σοβαρά τις προτάσεις τους, ότι τους ακούμε. Ε, αν υπάρχει δυνατότητα διαφορετικών απόψεων, ε, όντως ε, λαμβάνουμε υπόψη αυτές τις απόψεις που είναι φιλικές προς τους πολίτες και οι πολίτες συνειδητοποιούν ότι λαμβάνουμε υπόψη αυτά που προτείνουν και, δεν, και βρίσκουν ευήκοα ότα τέλος πάντων. Ε, η Επιτροπή Αναφορών θεωρεί ότι αυτό είναι επιτυχία και κρίμα ταυτόχρονα γιατί υπάρχει ένας σημαντικός κανόνας. Είμαι ο μόνος ε, ε, εισηγητής που έχει πολιτικά επιβιώσει από την πετή αυτή την επιτροπή. Δύο ε, άλλοι εισηγητές είχαν κάνει δύο πολύ σημαντικές προτάσεις να γίνονται οι ακρόασεις στο τέλος. Αυτό το φέραμε εμείς. Δεν θα ήταν στον κανονισμό αν εμείς δεν το είχαμε προτείνει. Επίσης, παλέψαμε ώστε η Επιτροπή Αναφορών να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτές τις ακροάσεις και σε αυτό δεν πετύχαμε σε επίπεδο αύκο όπως το θέλαμε τουλάχιστον. Παρ' όλα αυτά θα υπάρχει δυνατότητα για την Επιτροπή Αναφορών να εμπλακεί στις πρωτοβουλίες των πολιτών, επειδή ήταν ένας, ε, ανέφερε γίνεται με αυτού που δεν φτάνουν το 1 εκατομμύριο. Ε, όταν όμως ε, η Επιτροπή Αναφορών θέλει να συμμετέχει στην ακρόαση, μπορεί να κάνει αίτηση γι' αυτό και τα μέλη της Επιτροπής, οι συντονιστέ, συντονιστές, ε, πρόεδρος θα συμμετέχουν σε αυτή την, θα συμμετάσχουν σε αυτή την ακρόαση. Θα μας προσκαλούν δηλαδή ως Επιτροπή και θα μπορούμε καταλήλως να ε, εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία. Σας ευχαριστώ και σας ζητώ, σας προσκαλώ, όπως είπα και πριν, στο μέλλον να ασχοληθείτε με αυτές τις πρωτοβουλίες με τρόπο ανοιχτό το υποστηρικτικό και φιλικό προς τους πολίτες. Γιατί η Ευρώπη πρέπει να ακούσει τους πολίτες της και θέλει να ακούσει τους πολίτες της. Ε, αυτοί θα μας προτείνουν πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις αποφάσεις και τις πολιτικές μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφος Μπέκερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και για την ευκαιρία που μου δίνετε ε, να συζητήσουμε και να πούμε κάποιες σκέψεις μας ε, στον Επίτροπο της Κομισιόν. Μια σκέψη πολύ συγκεκριμένη, το γεγονός που ήδη αναγνωρίζεται, ότι έχουμε πολιτικά θεσμικά όργανα, όπως ε, είναι τα πολιτικά κόμματα, που αναφέρουν ε, ότι θέλουν αυτά τα όργανα, τις πρωτοβουλίες, να τα χρησιμοποιήσουν ε, ας πούμε, ο φόρος ε, στις συναλλαγές θεωρείται ως κάτι τέτοιο, ε, ως εργαλείο ε, που τα πολιτικά κόμματα έφεραν στο τραπέζι, ενώ στην πραγματικότητα συνέβη το αντίθετο. Είναι οι πολίτες που έφεραν το θέμα και είναι λίγο λαϊκίστικη αυτή η προσέγγιση. Θα ήθελα λοιπόν εμείς από το Κοινοβούλιο με την υποστήριξη της Κομισιόν, επειδή μπορείτε να επηρεάζετε τα μέσα την δημόσια, ε, τη, τη γνώμη, την κοινή γνώμη, να αναφέρετε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι σωστό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε τις παρεμβάσεις. Να δώσω το λόγο στον Επίτροπο Σάιφκοβιτς για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση της κυρίας Άουκεν για τα διάφορα ζητήματα που έφυξε. Πρώτον, την έκθεση που ετοιμάζει η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για την ε, χρηστή διαχείριση, χρηστή διοίκηση και φυσικά ε, παρακολουθούμε αυτή τη συζήτηση στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων πολύ στενά και ε, θεωρώ ο, μετά από την πρώτη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ότι δεν θα είναι πάρα πολύ εύκολο να χρησιμοποιηθεί ο γενικός κανόνας για διαφορετικές υποθέσεις. Αλλά ταυτόχρονα είναι προφανές ότι πρέπει όσο μπορούμε να βελτιώσουμε ε, την ποιότητα των, εργασιών μας, κυρίως ε, ε, προσανατολισμένη προς τις υπηρεσίες, διότι εμείς δουλεύουμε για τους πελίτες και επομένως πρέπει να υπηρετούμε τους πολίτες. Ε, πριν από μία εβδομάδα είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το θέμα αυτό με τον κύριο Διαμαντούρο, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, ο οποίος ε, κάνει και αυτός μία πρόταση για τις ε, χρηστές διοικητικές αρχές ε, και θεωρούμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό διότι ορισμένες φορές μπορούμε να επιτύχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα με ένα καλό κώδικα διοντολογίας που είναι καλύτερα συντονισμένο σε συγκεκριμένες προκλήσεις που αφορούν ε, τις συγκεκριμένες εργασίες μας ή ένα συγκεκριμένο τομέα και επομένως θα συνεργαστούμε και με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων αλλά και με τον διαμεσολαβητή πολύ στενά διότι εξετάζουμε και το ενδεχόμενο ε, να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την ε, ποιότητα της ε, ε διοίκησης. Ε, επίσης, επειδή είναι πολύ σημαντικό και το διαπίστωσα στη διάρκεια της συζήτησης, ε, ερωτικά να σας πω ότι στη συζήτηση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, όταν συζητούσαμε τον κανονισμό των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, ε, είδαμε πόσο μεγάλη σημασία δίνεται σε δεοντολογικά ζητήματα, σε δεοντολογικές αρχές, ε, πολιτικές ε, για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων και αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάποια από αυτά τα απαντήσαμε βελτιώνοντας τον κώδικα δεοντολογίας των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον οποίο επικαιροποιήσαμε πρόσφατα, ε, αλλά πάντα προσπαθούμε να δούμε τι μπορούμε να εισαγάγουμε, τι μπορούμε να βελτιώσουμε και τι μπορούμε να έχουμε στα πρότυπα για καλή διοίκηση και καλή συμπεριφορά των Ευρωπαίων ε, ε, υπαλλήλων. Όσον αφορά τώρα την οδηγία για το περιβάλλον και την αξιολόγηση αντικτύπου, αυτή είναι στη διαδικασία αναθεώρηση. Αυτή τη στιγμή είναι εξελίξει μια ευρύτατη δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πράγματι, σκοπεύουμε να κάνουμε πρόταση μέχρι το τέλο του έτου και ελπίζουμε πράγματι ότι η Επιτροπή σα ε, ή και εσεί ω μέλη τη Επιτροπή Αναφορών θα συνεισφέρετε προσωπικώς με τις ε, δικές σας τις ιδέες, ώστε να μπορέσουμε να τις ενσωματώσουμε στην πρόταση, να τις επεξεργαστούμε και θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο διότι θα μας βοηθήσει να κάνουμε μια επιτυχή αναθεώρηση της οδηγίας για την αξιολόγηση περιβαλλοντικού αντικτύπου. Αρκετά μέλη έθεσαν ε, την ερώτηση για τον 1049, την οδηγία 1049. Συμφωνώ ότι πολλές φορές τίθεται επιτάπητο στο ζήτημα αυτό και ξέρω ότι ε, το θέμα συζητήθηκε και στη διάρκεια της ακροασίας μου πριν από αρκετό καιρό όταν έγινε και χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτή τη στιγμή βλέπουμε κάποια θετικά βήματα και για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι αυτό που ήταν πάρα πολύ σημαντικό ήταν το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε σαφέστατα την άποψή του, αποφάσισε για το θέμα αυτό, το συζητήσαμε και με τη Δανική Προεδρία και ενημερωτικά να σας πω, η Δανική Προεδρία έχει υποβάλει ένα σχέδιο εντολή στην Κορεπέρ για να ξεκινήσει ε, ένας επίσημος ε, ε, γύρος συνομιλιών σε τριμερές επίπεδο για το θέμα αυτό. Θα συζητηθεί τη Δευτέρα και φαντάζομαι ότι πολύ σύντομα θα ξεκινήσει ο πρώτος τριμερής διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό είναι να δείξουμε ότι εμείς από πλευρά μας είμαστε καθόλου διατεθειμένοι να βρούμε λύσεις για το πώς μπορούμε να ε, έχουμε μια κοινή προσέγγιση, διότι νομίζω ότι το βασικό ζήτημα το οποίο μας διαιρούσε μέχρι τούδε ήταν ε, και είναι πάντα το ίδιο και προσπαθούμε να βρούμε λύση για να αντιμετωπίσουμε αυτό. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτή την εντός εισαγωγικών λισαβονοποίηση της πρόσβασης της πληροφορίας για τους πολίτες, διότι όπως γνωρίζετε μετά από την έναρξη ισχύω της συνθήκης της Λισαβόνας, η πρόσβαση στις πληροφορίες θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δεν ισχύει ακόμα αυτό και γι' αυτό ακριβώς ε, ε, προτείναμε ήδη από πέρσι να γίνει αυτή η μικρή αλλαγή ε, ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να χαίρουν των δικαιωμάτων τους και μετά να περάσουμε φυσικά στην πλήρη εφαρμογή. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να σεβαστούμε και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες επιπαραβάση και τους ε, τα θέματα ανταγωνισμού και το πώς ε, ε, μπορούμε να χειριζόμαστε εμπιστευτικέ και απόρριτες πληροφορίες. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ανήκυψε πολύ συχνά κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τότε βρήκαμε ένα καλό τρόπο για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτές τις εμπιστευτικές πληροφορίες και νομίζω ότι τώρα υπάρχει και μια καλή ε, ε, πρόοδος για το πώς μπορεί να γίνει αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ε, Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα υπάρχει ένα καλό μοντέλο που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία είναι πολύ ευαίσθητα βέβαια αν δεν κάνω λάθος και εκεί θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, να το σκεφτούμε ίσως λίγο περισσότερο. Ε, ο χαρακτηρισμός ας πούμε του κάθε εγγράφου διότι και για σας είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι πολύ σημαντικό και για μας να είμαστε βέβαιοι ότι όλα τα έγγραφα θα είναι διαθέσιμα μετά από κάποια πρώτη αίτηση. Ξέρετε ότι τώρα είναι πολύ μεγάλος ο όγκος των εγγράφων. Έχουμε ε, πάνω από 5.000 έγγραφα ετησίως. Υπάρχουν και κάποια έγγραφα τα οποία είναι και εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ε, εξετάζουμε πώς μπορούμε να επιλύσουμε όλες αυτές τις εκκρεμάτες με καλό τρόπο και αν υπάρξει συμφωνία νομίζω ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ε, καλά αποτελέσματα. Τώρα, όσον αφορά τη διαδικασία επιπαραβάση, ε, αρκετά μέλη ε, μου έθεσαν την ίδια ερώτηση, μπορώ να πω αφενός πρέπει να παραδεχτώ και ε, δεχτείτε αυτή την περιγραφή από πλευράς μου ότι εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρούμε ότι η παράβαση είναι μια μορφής αποτυχίας δικής μας. Δεν καταφέραμε δηλαδή ε, να επιτύχουμε τη μεταφορά της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ταυτόχρονα και με την ίδια ποιότητα σε όλα τα κράτη-μέλη και αυτή η διαδικασία επιπαραβάση είναι μιας μορφής διόρθωση. Ορισμένες φορές, ε, και φυσικά οι παραβάσεις είναι διαφόρων μορφών, ορισμένες φορές μπορεί να έχετε μια παρέμβαση ε, που δείχνει εσκεμμένη αδράνεια από πλευράς κρατών μελών και σε αυτή την περίπτωση δρούμε απευθείας ε, και όπως θα έχετε διαπιστώσει και από κάποιες πρόσφατες περιπτώσεις δεν διστάζουμε και να προσφύγουμε στα δικαστήρια κατά των κρατών μελών. Ε, σε κάποιε όμως περιπτώσεις είναι πολύ περίπλοκη νομοθεσία και εκεί δημιουργούνται προβλήματα, ιδίω σε κράτη-μέλη που έχουν ομοσπονδιακέ δομέ και χρειάζονται ε, ε, εκατοντάδε διαφορετικέ διαφορετικές νομοθετικές πράξεις για να γίνει η πραγματική μεταφορά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Και ταυτόχρονα κοιτάμε να δούμε πώς μπορούμε να συνδράμουμε τα κράτη-μέλη ώστε να γίνει κατάλληλη μεταφορά και κατάλληλη ε, εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας το συντομότερο δυνατόν, ώστε οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χαίρουν της ομοιομορφίας της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια και προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτό το χρόνο της διαδικασίας επιπαραβάσεις για να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε σωστή μεταφορά. Διότι όπως θα έχετε δει είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις οι οποίες φτάνουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θεωρούμε ότι αυτός είναι ο τρόπος που θα θέλαμε να συνεχίσουμε να ε, δραστηριοποιούμεθα και νομίζω ότι έτσι περιγράφει και το ζήτημα ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις διαδικασίες επί παραβάση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τώρα τον κύριο Γιάρ για τα ευρωπαϊκά σχολεία και συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Τα ευρωπαϊκά σχολεία είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Το έχουμε συζητήσει πολύ συχνά στο Σώμα των Επιτρέπων και όταν για ένα διάστημα ήμουν επίτροπος αρμόδιος για θέματα παιδείας, ε, το ότι ε, η ύλη ενός ε, ευρωπαϊκού σχολείου είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δημοσιεύεται. Δείχνει ότι υπάρχει υψηλή ποιότητα διδασκαλίας γλωσσών, ε, διδάσκονται οι ευρωπαϊκές αξίες, η ευρωπαϊκή ιστορία και εξηγείται γιατί είμαστε μαζί, τι πλεονεκτήματα υπάρχουν και τα παιδιά από τα ευρωπαϊκά σχολεία έχουν αυτά τα πολύ σημαντικά διαπολιτισμικά ωφέλη, τα οποία είναι δέλεα αργότερα και για τα πανεπιστήμια, αλλά και για τους ενδυνάμει εργοδότες τους. Και πρέπει να σας πω ότι προβληματίζομαι ιδιαίτερα, διότι αν δείτε τον προϋπολογισμό για τα ευρωπαϊκά σχολεία, ακόμα και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, δεν είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Αλλά φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου συζητάμε θέματα τα οποία νομίζω ότι σε πλήρης δημοσιονομικούς αριθμούς δεν είναι τόσο σημαντικά τα ποσά αυτά και νομίζω ότι θα αλλάξει η κατάσταση. Αυτό, αυτή η ευρωπαϊκή ύλη των ευρωπαϊκών σχολείων θα γίνει η κοινή γνώση και στα υπόλοιπα σχολεία. Θα μπορέσουμε να μοιραστούμε τη γνώση μας και την εμπειρογνωμοσύνη μας και να έχουμε σχολεία ε, τα οποία θα ε, μπορούν με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να λάβουν πιστοποίηση ότι διδάσκουν ευρωπαϊκά προγράμματα και ε, οι νέοι μαθητές θα μπορούν να λαμβάνουν ευρωπαϊκό απολυτήριο, κάτι το οποίο θα εκτιμούν ιδιαίτερα και τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, διότι θεωρείται ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Το τελευταίο συμβούλιο δεν ήταν πολύ ενθαρρυντικό επειδή όλα ε, τα κράτη-μέλη στο ε, Διοικητικό Συμβούλιο είπαν ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο επιμερισμό των δαπανών. Αλλά συγχρόνω είπαν ότι δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα. Οφείλω λοιπόν να ομολογήσω ότι όταν μιλάμε για τα ευρωπαϊκά σχολεία ανησυχώ κάπω και συνεπώ ε, προσπαθώ να έρθω σε επαφή απευθεία με τα κράτη-μέλη, με του πρέσβει, γιατί πρέπει να βρούμε μια σωστή λύση πάγια και για το μέλλον προκειμένου τα ευρωπαϊκά σχολεία να εξακολουθούν να λειτουργούν, να εξασφαλίσουμε την καλύτερη ποιότητα και να παρέχουν μια σωστή παιδεία για τους μαθητές. Τώρα, ως προς την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών πάλι, όπως είπαμε, αυτό θα δώσει νέο πολιτικό δυναμισμό ε, στις συζητήσεις μας ε, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι είδαμε ήδη με την άκτα που συζητήσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πώς η κοινή γνώμη μπορεί να κινητοποιηθεί μέσα από την κοινωνική δικτύωση, μέσα από αυτές τις διαδικασίες, πόσο πιο γρήγορα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα επίπεδα επικοινωνία για να εξηγήσουμε στους πολίτες ε, τι θέλουμε και νομίζω ότι αυτό θα μας αναγκάσει όλους όσοι εργαζόμαστε στον δημόσιο τομέα ε, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Επιτροπής ε, να ε, ενεργούμε πιο γρήγορα απέναντι στους πολίτες. Αλλά συγχρόνως αυτή η πρωτοβουλία νομίζω θα δώσει νέα δυναμική, θα εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες για ευρύτερες ευρωπαϊκές συζητήσεις προκειμένου τα ευρωπαϊκά θέματα να εξετάζονται όχι μόνο στο Στρασβούργο και στις αλλά και σε κάθε πρωτεύουσα και αυτό θα είναι πιο ενδιαφέρον για τους νέους, γιατί τότε θα αισθάνονται ότι πατώντα ένα κλικ με το ποντίκι τους μπορούν να στείλουν ένα μήνυμα ε, σε εκείνου που λαμβάνουν αποφάσει στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλε. Αυτό είναι σημαντικό να αισθάνονται ότι συμμετέχουν ε, στα κεκτενόμενα στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι ω προ το θέμα τη κυρία Κάν, δηλαδή τα, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία, τα Ευρωπαϊκά Σχολεία και επίσης αναφέρεται το θέμα της διαφάνειας και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη θαυμάσια συνεργασία που είχαμε όσον αφορά τη διαφάνεια. Πρόσφατα περάσαμε 5.000 μονάδων που έχουν εγγραφεί σε αυτό το κατάλογο της διαφάνειας, δηλαδή πολλά άτομα βλέπουμε λοιπόν μια θετική πίεση που ασκείται για στις οργανώσεις, ε, στους θεσμούς, σε φορείς, ε, σε δικηγορικά γραφεία, σε επιχειρήσεις, ε, να εγγραφούν σε αυτό τον κατάλογο διαφάνειας. Και αυτό έχει σημαντικές συνέπειες, διότι βλέπουμε πώς όλες αυτές οι μονάδες, όλοι αυτοί οι φορείς αυξάνονται και νομίζω ότι ε, το γεγονός ότι έχουμε ένα τόσο μεγάλο αριθμό ε, εγγεγραμμένων είναι πολύ σημαντική και ευχαριστούμε ε, τη συνεργασία, για τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Τώρα ελπίζουμε ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο, το, συμβούλιο, το δικό μας Συμβούλιο θα βρίσκεται υπό μορφή παρατηρητών και θα στείλουμε ένα πολύ θετικό σινιάλο και στον τομέα της διαφάνειας. Ο κ. Χέφνερ ανέφερε ότι ένα καλό ξεκίνημα είναι σημαντικό, αλλά πιο σημαντικό θα είναι πώς θα διαχειριστούμε την πρωτοβουλία στους Ευρωπαίους πολίτες στο μέλλον. Και αυτό θα είναι κάτι σημαντικό για όλους μας. Θα μάθουμε από αυτά. Και το πρώτο τεστ θα γίνει όταν έχουμε ένα εκατομμύριο υπογραφές, όταν δοκιμάσουμε την υποδομή που υπάρχει σε κάθε χώρα μέλος για να δούμε αν όλα λειτουργούν ομαλά όπως μας έχει αναφερθεί και πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη φάση, την ακρόαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο και είμαι βέβαιος ότι θα βρείτε μία ε, μέθοδο να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα και εμείς ε, πώς από την Επιτροπή θα επικοινωνήσουμε, ε, πώς θα εξηγήσουμε γιατί υιοθετήσαμε αυτή έναντι της άλλης απόφαση διότι ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε την πρώτη περίπτωση θα είναι ένας σαφής δείκτης προς τους πολίτες, για να δουν με πόση σοβαρότητα ε, αντιμετωπίζουμε το θέμα, ώστε και οι πολίτες να καταλάβουν ότι αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα. Τώρα, προς ενημέρωσή σας σχετικά με την επεξεργασία όλων αυτών των θεμάτων από τα διάφορα κράτη-μέλη, ε, συγκροτήσαμε μια ομάδα εργασία εμπειρογνωμόνων που θα είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των θεμάτων τη πρωτοβουλία αυτή στα κράτη-μέλη και γίνεται ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών και των θεμάτων που είναι σημαντικά για την κράτη-μέλη. Και αυτό όμω μα βοηθάει να επιταχύνουμε την διαδικασία προετοιμασία ώστε να υπάρχει ετοιμότητα από όλα τα κράτη-μέλη. Τώρα, το τελευταίο θέμα του κύριου Μπέκερ. Θα θυμάστε ότι ήταν ένα από τα θέματα τα οποία συζητήθηκε διαμακρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισαν ότι μόνο οι πολίτες μπορούν να συγκροτήσουν την Επιτροπή των Πολιτών. Είναι λοιπόν απόλυτα φυσιολογικό αυτό το θέμα να ε, αφορά τους πολίτες. Και το θέμα είναι πώς θα κατορθώσουν να επιτύχουν ε, την υποστήριξη για αυτή την πρωτοβουλία του Ευρωπαίου Πολίτη. Και συμφωνώ με την κυρία Μαντσόνη που είχε γράψει πρόσφατα ένα πολύ καλό άρθρο για αυτό το θέμα και είχε πει πολύ σωστά ότι το 1 εκατομμύριο πολίτες είναι ένας αριθμός πολύ σημαντικός. Ε, πρέπει να το λάβουμε υπόψη σοβαρά και το να φτάσει κανείς στο 1 εκατομμύριο πολίτε είναι καλύτερη ε, δικλίδα ασφαλείας για οποιαδήποτε ολίσθηση. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Σεύκοβιτς. Σας ευχαριστώ πολύ που μας δώσετε αυτή τη δυνατότητα και εμείς φυσικά θα φυλάξουμε ως ε, θησαυρό αυτό το ε, άνοιγμα που κάνατε για συνεργασία και θα φροντίσουμε ε, να νομιλούμε με τον κύριο Σεύκοβιτς για όλα τα θέματα που μας ανεσχυνούν και για το θέμα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών αλλά και για όλα τα υπόλοιπα θέματα που είναι αρμοδιότητα του Αντιπροέδρου Σεύκοβιτς. Σας ευχαριστώ και πάλι για το γεγονός ότι είστε τόσο διαθέσιμος. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Αναφορά 197 του 2012, όπως αποφασίσαμε σήμερα το πρωί, τροποποιώντας την ημερήσια διάταξη, την ε, Αναφορά λοιπόν του κυρίου Φραντσέσκο Σαλτίνη για το σχεδιαζόμενο χώρο υγειονομική ταφή αποβλήτων κοντά στη Ρώμη, στο Κόρκολε, στο Λάτσιο. Είναι παρόντες ε, για την αναφορά δύο από τους υπογράφοντες της αναφοράς. Ο πρώτος, ε, στον οποίο θα δώσω το λόγο για πέντε λεπτά, είναι ο κύριος Φραντσέσκο Σαλτίνη, εκπρόσωπος της ε, Επιτροπής Μηδενικά Απόβληπτα του Κορκόλε. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους τους ε, βουλευτές που είναι παρόντες που μας έδωσαν τη δυνατότητα να σας ε, παρουσιάσουμε ε, την άποψή μας εδώ στο Κοινοβούλιο. Έχουμε έρθει εδώ για να σας παρουσιάσουμε ένα πρόβλημα το οποίο δεν αφορά μόνο τη δική μας την περιοχή ή μάλλον δεν σας το παρουσιάζουμε εμείς μόνο γιατί αφορά μόνο εμάς την περιοχή μας αλλά γιατί θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο είναι λίγο πολύ γενικευμένο σε όλη την ε, περιοχή της ε, ε, ε αλλά κυρίως και στη δική μας την περιοχή είναι ένα πρόβλημα και περιβαλλοντικό αλλά και ε, οικονομικό και θα το δούμε στην ε, πορεία. Σήμερα δεν είναι πολύ εύκολο να κατανοήσουμε προς ποια κατεύθυνση κινείται αυτή η ανάγκη να λυθεί το πρόβλημα από πλευράς ε, τοπικών αρχών. Το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων, το οποίο δεν το διαχειριζόμαστε και με τον καλύτερο τρόπο. Από την τελευταία παρέμβαση του Υπουργού Περιβάλλοντος στην Ιταλία, ο οποίος προσφέρει ουσιαστικά τα μέσα προκειμένου να μπορέσουμε να διαφύγουμε από αυτό το φαύλο κύκλο της διαχείρισης των αποβλήπτων, δηλαδή με αυτό τον τρόπο ε, δεν ε, ε, διευκρίνησε την κατάσταση, δεν μας εξήγησε πολύ καλά πού θα καταλήξουμε με όλη αυτή την υπόθεση. Τα βασικά ζητήματα που μας ενδιαφέρουν, δηλαδή οι, οι, οι αρχές φαίνεται να είναι όλο ένα και πιο διατεθειμένες να μην προσπαθήσουν να φύγουν, διότι τα μέσα τα οποία προτείνει ο υπουργό κλείνει δεν γίνονται αποδεκτά, ε, πάντα κάτι πηγαίνει στραβά και ε, η κατάσταση Ε, κανονικά θα έπρεπε να είναι δεχτή. Να δεχτούμε αυτό που προτείνει ο Υπουργό και να ε, προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Εν μέσω λοιπόν όλων αυτών των διαφορών μεταξύ του Υπουργού και το, της τοπικής αυτοδιοίκησης βρισκόμαστε εμείς, δηλαδή αυτοί που ζούμε στην περιοχή, οι κάτοικοι και ε, το θέμα αυτό που αφορά εμάς πιο συγκεκριμένα ε, μας απασχολεί εδώ και ένα χρόνο, δεν γνωρίζουμε ε, ποιο θα είναι το μέλλον μας, ζούμε ένα εφιάλτη και μπορεί να βρεθούμε με μια χωματερή 500 μέτρα από το σπίτι μας. ουσιαστικά έχουμε μια δαμόκλειο σπάθη που επικρέμεται πάνω από το κεφάλι μας και μας λέει ότι δεν είναι τίποτα ε, σαφές και αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο ε, διότι ε, θεωρείται ότι δεν είναι κατεπίγουσα η ανάγκη, στην ε, πραγματικότητα δεν υπάρχει. Το είπε επανειλημμένος ο Υπουργός, δεν υπάρχει κάτι κατεπήγον. Ε, ο Υπουργός ε, μέσα στα συνήθη σχέδιό του ετοίμασε ένα πρόγραμμα για να λύσουμε την κατάσταση και αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει κατεπίγουσα κατάσταση για μας. Στο όνομα λοιπόν αυτού του κατεπήγοντος δεν μπορούμε να μη σεβαστούμε τους κανόνες και την ομοθεσία η οποία εκπονήθηκε ακριβώς για να υπάρχουν δεσμεύσεις για τα θέματα αυτά. Δεν μπορούμε να ζητάμε από τους πολίτες να αναλαμβάνουν την ευθύνη τους ε, και ε, να είναι νόμιμοι όταν δεν γίνονται αποδεκτά από την ίδια την κυβέρνηση αυτά τα θέματα. Ε, προσπαθούμε ε, με εξαιρετικές εξουσίες να ξεπεράσουμε κάποιες δεσμεύσεις και κάποιους κανόνες, οι οποίες κατά την άποψή μου δεν είναι ακριβώς νόμιμες. Ζητάμε από τους πολίτες... Ε, ε, να ε, κάνουν κάτι και δεν γίνεται αποδεκτή για συζήτηση. Το να έρθουν οι πολίτε σε μία συνάντηση όμως δεν σημαίνει ότι νομιμοποιείται μια κατάσταση. Αυτό τον εφιάλτη ζούμε, με αυτό το άγχος ζούμε καθημερινά. Δεν έχει εφιαλτη ζουμε με αυτο το αγχο τίποτα ε, για να... Ε, λύσουμε αυτό το θέμα του κατεπήγοντος το οποίο ε, επικαλούνται οι τοπικές αρχές ε, και για την ανικανότητά τους ε, για το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων διότι κατά την άποψή μας είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων. Η περιοχή του Λάτσιο και η περιφέρεια ε, χρησιμοποιεί ωραία λόγια, χρησιμοποιεί συνέχεια διάφορους κανονισμούς οποίες επικαλείται για τη διαχείριση των αποβλήτων και μετά για όλα αυτά ε, δεν καταφέρνουν να εγκρίνουν τίποτα και μένουμε όπως είναι η κατάσταση χωρίς να αλλάζει τίποτα. Χρησιμοποιούνται λοιπόν ε, οι για να διαχειριστούμε την, ε, ε, τα απόβλητα. Και οι πολίτες δεν μπορούν να ζουν πλέον με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορεί να είναι πια αυτός ο δρόμος, διότι πρόκειται για ένα φαύλο κύκλο, τον οποίο υποχρεώθηκαν να ακολουθήσουν από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα απόβλητα όλα αυτά τα χρόνια και φυσικά πληρώνουν και τις συνέπειες και από τις ε, ε, ε παρατάσεις που γίνονται στις εξαιρέσεις αυτές και από το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται σχεδόν υποχρεωτικά αυτές οι χωματερές. Δεν υπάρχει άλλο σύστημα και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο αυτό, διότι δεν υπάρχουν άλλοι. Είναι αδύνατο να αλλάξει το σύστημα της διαχείρισης των αποβλήτων, αλλά αυτό αποδείχθηκε ότι δεν είναι αλήθεια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ζητάει να πληρώσουμε γιατί είμαστε παράνομοι. Εξακολουθούμε να είμαστε παράνομοι και παρόλα αυτά εξακολουθούμε να επιμένουμε να φτιάξουμε μια χωματερή σε περιοχές τις οποίες είναι αδύνατο να δημιουργηθεί χωματερή λόγω εδαφικών, περιβαλλοντικών, υδρογεολογικών ε, ε, προσκομμάτων και ελοχεύει ο κίνδυνος να γίνει μια τεράστια ρήπανση και της περιοχής αλλά και του αέρα και του νερού της περιοχής. Οι πολίτες είναι έτοιμοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους αλλά ζητούν Ζητώ συγγνώμη, με κρυγορό. Ζητούν λοιπόν να τους εκπροσωπήσει κάποιος ο οποίος θα μπορέσει να λάβει υπόψη τις θέσεις των πολιτών και να μας συνοδεύσει κάποιος σε όλη αυτή την πορεία ώστε πραγματικά να φτάσουμε σε μια νόμιμη κατάσταση. Αυτό ζητάμε από την Επιτροπή σας. Δεν μπορείτε να δηλητηριάσετε μια περιοχή και δεν μπορείτε να δηλητηριάσετε τους πολίτες στο όνομα μιας κατεπίγουσας κατάστασης που δεν υπάρχει. Σας ευχαριστώ και τώρα να δώσουμε το λίγο ε, στον κύριο Μαρτίνο τον Ιμιέλε ο οποίος είναι από την Επιτροπή της ε, Γειτονιάς να ευχαριστήσω και πάλι τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών και να ευχαριστήσω ε, και τους εκπροσώπους ε, της τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι εδώ. Θα σας διαβάσω ε, τι περιείχε αναφορά μου. Σα ευχαριστώ για την προσεκτική συνεργασία που μου έδωσε τη δυνατότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωσης να διεκδικήσουμε ένα δικαίωμα ε, για τη διατήρηση μια περιοχή που είναι πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Απελείται ένα αρχαιολογικό αγαθό το οποίο ανήκει στην πολιτιστική ε, κληρονομιά. Είναι η διά, διάσημη βίλα του Ανδριανού που βρίσκεται σε μια εξαιρετική κατάσταση σε σχέση με αντίστοιχα αρχαιολογικά μνημεία και οι ε, οσμές από την χωματερή, εάν κατασκευαστεί, κατά πάσα πιθανότητα ε, σημαίνουν ότι θα πάψει να είναι αυτός ο αρχαιολογικός χώρος ε, ως πολιτιστικό μνημείο της ανθρωπότητας. Μάλιστα η UNESCO διαβίβασε ότι ξεκίνησε μία διαδικασία επιτήρησης από τον Ιούνιο ε, θα ξεκινήσει μάλλον τον Ιούνιο σε περίπτωση που δημιουργηθεί η χωματερή αυτός ο χώρος, εάν ε, κατασκευαστεί όντως, θα βρίσκεται στα 300 μέτρα από τη βίλα του Ανδριανού και 100 μέτρα από την περιοχή προστασίας της βίλας του Ανδριανού. Σήμερα, χάρη στην παρέμβαση του Υπουργού Κλίνη, που είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος της Ιταλίας, αυτή η υπόθεση της χωματερής ε, στην περιοχή της βίλας του Ανδριανού φαίνεται ότι θα σταματήσει και χάρη από την αναγνώριση ε, περιβαλλοντικών δεσμεύσεων... το Υπουργείο υποστηρίζει ότι μάλλον είναι αδύνατο να εγκατασταθεί στην περιοχή αυτή η ε, χωματερή. Και διευκρινίζει ότι τα χαρακτηριστικά του εδάφους είναι κατώτερη κατά τρεις βαθμούς ε, ε, όσον αφορά τη διαπερετότητα που καθορίζεται με τη συγκεκριμένη νομοθεσία για τα θέματα αυτά, δηλαδή τη μεταφορά της οδηγίας 2060 ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Για να σας εξηγήσω λίγο τι γίνεται και χρησιμοποιώ κάποιους ιταλικούς όρους, αναφερόμαστε σε μια ιστορική τοποθεσία και πρέπει να πούμε ότι η ιστορία προέρχεται από τον ελληνικό όρο ιστορία ε, και σημαίνει ότι είναι ιερή, σημαίνει γνώση που οδηγεί στη γνώση, σημαίνει ότι βλέπω, ενημερώνομαι, γνωρίζω, ερευνώ και όλοι αυτοί είναι παράγοντες οι οποίοι ε, διαβάζονται καθημερινά από την ευρωπαϊκή κοινότητα και στα θέματα του περιβάλλοντος και των αποβλήτων το κάνει με την οδηγία 1997-11, 1997-31, ε, καθώς επίσης και την οδηγία για τη διαχείριση των υδάτων. Και επίσης βλέπουμε και τι γίνεται με την διαχείριση των αποβλήτων και με ε, τα όσα μπορούμε να έχουμε εν είδη εξαίρεσης ε, ως κατεπίγουσα κατάσταση. Και φαίνεται ότι όλα αυτά διαψεύδουν αυτές τις υποδείξεις. το περιβάλλον είναι ένα αμάλγαμα παραγόντων είναι εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη ζωή μας. Είναι οι φυσικοί παράγοντες, το έδαφος, το νερό, η ατμόσφαιρα, η πανίδα, η χλωρίνα, οι οικονομικοί, οι κοινωνικοί παράγοντες, ε, παράγοντες που βοηθούν την υγεία, ιστορικοί και επιστημονικοί που επηρεάζουν τη ζωή μας καθημερινά. Όταν αναφερόμαστε λοιπόν σε μία χωματήρη, δεν θα πρέπει να γίνεται μία αξιολόγηση και μία συζήτηση μεταξύ ενός Υπουργείου και ενός Επιτρόπου αρμόδιου για τα θέματα αυτά, αλλά και μέσω αντιπροσωπιών των πολιτών που εκπροσωπούν αφορούν ε, τους τη της περιοχής, γιατί αυτοί ζουν σε μια περιοχή, είναι αυτοί που μπορεί να υποστούν οικονομικέ και κοινωνικέ συνέπειε στη συνέχεια και ε, θα μπορούν να, μπορεί να ζουν και στην ανασφάλεια και να είναι και επικίνδυνη η καθημερινή του διαβίωση και υγεία. Αυτά άλλωστε λέει και ο Παγκόσμιο Οργανισμό τη Υγεία. Δηλαδή, ε, δεν χρειάζεται να υπάρχει μόνο έλλειψη ασθένεια, αλλά θα πρέπει και να υπάρχει και μια γενικότερη ευημερία ε, σκεφτείτε την αρχική έκταση. Αναφερθήκανε στα τέσσερα στρέμματα. Ο Επίτροπος ε, μίλησε για περίπου 164 ε, στρέμματα, 164 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και για την περιοχή του Τίβολη σημαίνει ότι εκτινόμαστε σε μια περιοχή 68 τετραγωνικών χιλιόμετρων και όλα αυτά κοντά σε αρχαιολογικούς χώρους ή και πάνω σε αρχαιολογικούς χώρους και σε μια περιοχή στην οποία ε, φτάνουν τα ύδατα τα από εκεί και πέρα ε, τη χάνουν επεξεργασίες και χρησιμοποιούνται ε, από την εταιρεία υδάτων για την χρήση πόσιμου και νερού για την υδροδότηση μιας μεγάλης περιοχής της Ρώμης και πρέπει να πούμε και ότι σε εκείνη την περιοχή υπάρχουν και πηγάδια διότι εκεί δεν υπάρχει ε, κατάλληλη υδροδότηση σε κάποιες περιπτώσεις γιατί είναι μεγάλη απόσταση και ήδη εκ των προτέρων λαμβάνουν και πόσιμο νερό από πηγάδια τα οποία μπορεί και να είναι μολυσμένα ε, και δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι και σε μικρή απόσταση περνάει και το υδραγωγείο ε, της Άκουα Λαμάτσα το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό. Τα όσα σκοπεύει να κάνει ο Υπουργό Κλίνη για την περιοχή αυτή μας φαίνονται πάρα πολύ καλό και εμείς ουσιαστικά ζητάμε τη βοήθεια και την παρέμβαση της Επιτροπής σας ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν όσα είπε ο Υπουργό και να μπορέσουμε σε σχέση με την καθυστέρηση η οποία έχει γίνει ήδη στην περιοχή του Λάτσιο να δοθεί μια ετήσια παράταση ε, με βάση τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Μόνο με τη βοήθειά σας νομίζω ότι μπορούμε να ε, ξεχάσουμε αυτή την άθλια ιδέα ε, για τη διαχείριση των αποβλήτων και τα λάθη τα οποία ε, θα έχουν υπόφθηνη για την υγεία και την ασφάλειά μας ε, στην περιοχή αυτή που είναι και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η αξία της περιοχής αυτής, που επαναλαμβάνω ότι ανήκει και στην πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μανκανάρο, εξ Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Sì, buongiorno. Ehm, dunque, la... Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί πάρα πολύ στενά το θέμα της διαχείρισης των αποκλήτων στην περιοχή του Λάτσιο. Είναι ένα περίπλοκο ζήτημα για το οποίο ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και χρόνια. Έχουν ξεκινήσει ήδη δύο διαδικασίες επί παραβάση, οι οποίες είναι εξελίξει και αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων στην περιοχή του Λάτσιο. Και προσφάτως ξεκίνησε και μία νέα έρευνα που αφορά ε, πολύ συγκεκριμένα τη διαχείριση της περιοχής ε, της Μαλαγκρότα. Ε, εξ όσων ανακοινώθηκε θα κλείσει η χωματερή της Μαλαγκρότα και από εκεί και πέρα βλέπουμε τι θα γίνει και τι μέτρα θα εγκρίνουν οι Ιταλικές αρχές για να υπάρχει σωστή διαχείριση των αποβλήτων ε, της περιοχής. Αυτό φυσικά είναι και το αντικείμενο της αναφοράς που συζητούμε αυτή τη στιγμή. Και θα πρέπει να σας πω ότι στις τελευταίες εβδομάδες και τους τελευταίους μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε αρκετές καταγγελίες και υποδείξεις ε, που αφορούν το κατά πόσον θα δημιουργηθούν χωματερές στην περιοχή του Λάτσιο για το τι θα γίνει μετά το κλείσιμο της Μαλαγκρότα που είναι η βασική χωματερή της πόλης. Βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να λάβει θέση για το κατά πόσον πρέπει ή δεν πρέπει να γίνονται χωματερές ή άλλες ε, εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων στην τάδε ή στη δίνα περιοχής. Αλλά αυτό το οποίο τέθηκε υπόψη της Επιτροπής είναι ότι Υπάρχει διάταγμα του Υπουργείου, ε, του Συμβουλίου Υπουργών ε, του Σεπτεμβρίου του 2011 για την καταπήγουσα διαχείριση των αποβλήτων ε, της Ρώμης, η οποία μπορεί να έχει παρέκκληση για μια σειρά από κανόνες, κυρίως του περιβαλλοντικού κώδικα και κάποιων κανόνων που αφορούν τα θέματα της αξιολόγησης περιβαλλοντικού αντικτύπου και της στρατηγικής περιβαλλοντικής αξιολόγησης. Πρόκειται λοιπόν για θέματα που αφορούν κυρίως ε, την ε, διαβούλευση των πολιτών, στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας ε, αξιολόγησης και των πιθανών επιπτώσεων που μπορούν να έχουν τα διάφορα περιβαλλοντικά σχέδια, τα οποία πρέπει να γίνουν πριν δοθεί έγκριση για οποιοδήποτε πρόγραμμα υποδομών το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ε, των ε, εν λόγω οδηγών, ε, οδηγιών, κυρίως για τη διαχείριση των αποβλήτων. Εδώ έχουμε σχέδιο υποδομών που εντάσσονται στο σχέδιο εφαρμογής της οδηγίας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν στα πλαίσια της έρευνάς της και μιας επιτόπου έρευνας που ίσως γίνει, αυτό θα το δούμε, θα ζητήσει διευκρινήσεις από τις Ιταλικές Αρχές και ούτως ή άλλως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στείλει και μια γραπτή κοινοποίηση για το τι μέλη γενέστε με αυτή την αναφορά σε επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Ε, η κατάσταση είναι υπό εξέταση αυτή τη στιγμή από πλευράς Επιτροπής ε, από τα όσα ακούσαμε. Είναι εδώ σήμερα και κάποιοι εκπρόσωποι των ε, τοπικών αρχών από πλευράς Ιταλίας που ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό υπάρχει ο Επίτροπος Εκτάκτων Θεμάτων, ο Τζουζάπε Καταρόρε, έχουμε και τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω τώρα το λόγο στους δύο κυρίους και να ξεκινήσουμε με τον κύριο Πεκοράρο. Ευχαριστώ. Χαιρετώ τα μέλη της Επιτροπής, χαιρετώ και τους πολίτες ε, που ε, κατέθεσαν αυτή την αναφορά. Καταρχάς, πρέπει να πω ότι εγώ ε, δέχτηκα αρκετές επιτροπές από τότε που ανέλαβα καθήκοντα στις αρχές Σεπτεμβρίου και αυτές οι επιτροπές των πολιτών μέχρι ε, τα μέσα του Νοεμβρίου ήταν αυτές που δέχτηκα. Δεν ξέρω αν οι παρόντες ήταν ε, σε αυτές τις επιτροπές ή εγώ δέχτηκα κάποιους άλλους αλλά τέλος πάντων εγώ είδα αρκετούς εκπροσώπους πολιτών. Είχα και έχω συνεχείς επαφές με τις ε, τοπικές αρχές και με ε, τις αρμόδιες υπηρεσίες της κυβέρνησης που ασχολούνται με τα θέματα των αποβλήτων. Και κατόπιν λάβαμε υπόψη τις διάφορες παρατηρήσεις και τα στοιχεία που λάβαμε από τους πολίτες. Ένα από τα πράγματα που ε, ακούστηκαν είναι ότι ε, δεν υπήρξε κάποια ε, παράβαση. το θέμα αυτό της, του κλεισίματος της κομματορής αποφασίστηκε από την κυβέρνηση το 2011 διότι υπήρχε πρόβλημα και έπρεπε να υπάρχει μια διαχείριση αποβλήτων που θα τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και θα είναι και σύνομο ως προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για να υλοποιηθεί λοιπόν αυτό το σχέδιο, σύμφωνα με την κυβέρνηση και με τις τοπικές αρχές, έπρεπε να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος για να γίνουν τα απαραίτητα έργα. Η μεταβατική περίοδος η οποία θεωρείται εκτάκτου χαρακτήρα, αλλά είναι και εκτάκτου χαρακτήρα διότι αναλαμβάνει το θέμα αυτό κάποιος ο οποίος δεν είναι αρμόδιος ε, για θέματα αποβλήτων και έχει συγκεκριμένες εξουσίες, μεταξύ των οποίων και να ε, εντοπίσει πού θα μπορούσαμε να έχουμε χωματερές. Και φυσικά όλα αυτά για να μπορέσει να υλοποιηθεί το σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων, το οποίο έχει ήδη παρουσιάσει η περιοχή του Λάτσιο και έχει ήδη ε, υποβληθεί στις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές. Για να μπορέσουμε λοιπόν να ξεπεράσουμε αυτή τη μεταβατική περίοδο από πλευράς μου και από πλευρά συνεργατών μου αναλάβαμε ε, να βρούμε, όπως σας είπα, κάποιες περιοχές οι οποίες προτάθηκαν από την περιοχή του Λάτσιο, ε, έγιναν ε, πολύ σημαντικές έρευνες από πλευρά συμβούλων και φυσικά ε, το εξέτασαν και ε, διοικητικές αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για αυτά τα θέματα. Έγιναν κάποιες επιλογές Και είναι προφανώ ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποιε επικρίσει για αυτέ τι περιοχέ. ε, και εγώ επανειλημμένω έχω πει ότι δυστυχώ η Ρώμη αυτή τη στιγμή δεν έχει ευνοϊκές συνθήκες για να μπορέσει να κάνει κάποιες ε, επιλογές τις οποίες θα βρίσκουν όλες, όλοι ε, κατάλληλες και θα συμφωνούν απαραίτητο και πολίτες όσον αφορά ε, την ομοθεσία και για τον ομάρχη και από πλευράς ε, των συνεργατών μου. Εγώ πρέπει να πω ότι αρνούμε τις παρατηρήσεις που έγιναν, όπως επίσης απορρίπτω και οτιδήποτε γίνεται και εμείς θεωρούμε ότι μπορούν να οδηγήσουν σε ρήπανση ε, του αέρα και των υδάτων. Διότι ακριβώς ε, και ως έκτακτος επίτροπος, διότι εγώ δεν είμαι αρμόδιος για τα θέματα αυτά, Και ο έκτακτος αυτός χαρακτήρας μου προβλέπει ότι η δική μου υποχρέωση είναι ε, η διαχείριση των αστικών λιμάτων. και όταν μιλάμε για αστικά απόβλητα θα πρέπει να ε, υπάρχει και συνέπεια προς την ισχύουσα νομοθεσία για το θέμα αυτό. Και η νομοθεσία προβλέπει ο νομάρχης ή μάλλον η νομαρχία για να το πω καλύτερα να μπορεί να βρει και να ε, ε, προβλέπει χώρους υγειονομικής ταφής των αποβλήτων για την επεξεργασία των αστικών αποβλήτων και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Έχουν γίνει αρκετές συνεδριάσεις για να αυξηθεί ο αριθμός των συσκευών αυτών ε, στην ε, περιοχή του Λάτσιο. Αυτή τη στιγμή έχουμε τέσσερις συσκευές ε, δεν λειτουργούν όλες σε πλήρως καθεστώ, αλλά ελπίζουμε να μπορέσει να γίνει αυτό το συντομότερο και είμαστε υπέρ και της υλοποίησης ενός πέμπτου ε, τέτοιου χώρου κοντά στην ε, πόλη της Ρώμης. Και αυτό φυσικά θα ε, δούμε και κατά πόσον θα μπορούμε ε, να έχουμε και απόβλητα τα οποία δεν θα είναι ως μοιρά και θα υπάρχει και απόλυτη επεξεργασία τους. Διότι ε, διαφορετικά απόβλητα ε, θα ήταν παράνομο ούτως ή άλλως ε, και θα ήταν και ενάντια στην ισχύουσα νομοθεσία και την Ιταλική αλλά και την Ευρωπαϊκή. Δεν ξέρω κυρία Πρόεδρε αν μπορώ να συνεχίσω. Έχω πέντε λεπτά ή... Κοιτάξτε, δεν έχετε άλλο χρόνο. Αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, σα ακούμε πολύ σύντομα, διότι πρέπει να δώσουμε το λόγο και στου υπολείπου. Δύο στοιχεία πολύ σύντομα. Καταρχά, η βίλα του Ανδριανού βρίσκεται 2.400 μέτρα από τη χωματερή που θα κατασκευαστεί και από την χωματερή του Κορκόλε, πιθανή χωματερή του Κορκόλε και τη βίλα του Ανδριανού υπάρχει ένας αυτοκινητόδρομος ενδιάμεσα και νομίζω ότι από περιβαλλοντική σκοπιά ε, αυτό είναι πιο σημαντικό από μια χωματερή η οποία θα χρησιμοποιηθεί μόνο για μια προκαθορισμένη διάρκεια 2-2,5 ετών. Δεν θα ε, ξεπεράσουμε αυτή τη διάρκεια. Όσον αφορά τώρα τα στρέμματα, εμένα δεν μου βγαίνουν τα 160 στρέμματα που λέτε εσείς. Είναι πολύ λιγότερα. Ε, είμαστε στα 10 στρέμματα έκτασης και μόνον ε, για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις χωματερές. Τα 160 στρέμματα αφορούν όλη την περιοχή, αλλά φυσικά δεν μας ενδιαφέρει εμάς όλη η περιοχή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βεσέλη εξ ονόματος της ε, περιφέρειας, αν θέλει να προσθέσει κάτι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ και σας και όλους όσους είναι παρέντε. Η νομαρχία της Ρώμης ε, για το θέμα αυτό της χωματερής του Κορκόλε ασχολήθηκε και για τις υπηρεσίες που προτείνει η περιοχή του Λάτσιο και έπρεπε να εγκρίνει ένα προκαταρκτικό σχέδιο αυτής της ε, περιοχής ώστε να μπορέσει να γίνει μία προσωρινή χωματερή για τις ε, εγκαταστάσεις ε, υγειονομικής ταφής αποβλήτων που υπάρχουν στην Ομαρχία της Ρώμης. Μας ενδιαφέρει κυρίως η ε, περιβαλλοντική προστασία και ο σεβασμός της οδηγίας για τη διαχείριση των αποβλήτων ε, και βάσει της Ιταλικής νομοθεσίας που μεταφέρει αρκετές ευρωπαϊκές οδηγίες και μπορέσαμε ε, στη συγκεκριμένη περιοχή να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν κάποια βασικά στοιχεία που αφορούν το προκαταρκτικό σχέδιο που προτείνει η περιφέρεια και αναφέρονταν πιο συγκεκριμένα στην ελληπή τεκμηρίωση και σε κάποια στοιχεία τα οποία κατά την άποψή μας θα πρέπει να εμβαθύνουμε περισσότερο, ιδίω όσον αφορά ε, τα ε, υπόγεια αλλά και η υπέρχεια ύδατα, αλλά και το γεγονός ότι υπάρχουν ε, προσκόμματα και από περιβαλλοντική σκοπιά αλλά και λόγω της, του γενικότερου χωροταξικού σχεδίου της νομαρχίας της Ρώμης, όπου διαπιστώνεται ότι σε αυτή την περιοχή υπάρχουν ε, ε πρωτογενή υδρολογικά δίκτυα τα οποία είναι υψή τη σημασίας και δεν θα πρέπει να υπάρξει χώρος αποβλήτων διότι αυτό θα ήταν εις και κάποιων αρχών που αφορούν την προστασία της βιοποικιλότητας. Δηλαδή, ε, βάσει αυτών των επιχειρημάτων και κυρίως από τα όσα ε, έγιναν ε, ως προκαταρκτική αξιολόγηση σε αυτό το προκαταρκτικό σχέδιο που παρουσιάστηκε, η περιοχή της Ρώμης είχε αναφέρει ότι ήταν απαραίτητο και διαπιστώσει ότι ήταν απαραίτητο να εμβαθύνουμε περισσότερο κυρίως ε, για τα στοιχεία που δίνονται για, μέσω μιας ε, υδρογεωλογικής μελέτης, ώστε να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε αν ε, όντως ε, τεχνικός είναι ε, εφικτό να υπάρχει αυτό το σύστημα για τη συλλογή των υδάτων και θα πρέπει να γίνει μια πιο εις μελέτη της τοπικής υδρογεωλογίας για να μπορέσουμε να δούμε αν μπορέσουμε να έχουμε και σωστή παρακολούθηση της χλωρίδας και της πανίδας και να δούμε και τι γίνεται από εκεί και πέρα και για τον υδροφόρο ορίζωσης και για να δούμε κατά πόσον ξεπερνάτε αυτό το θέμα της ασφάλειας. Πέρα από αυτές τις τεχνικές ε, συζητήσεις, η ε, νομαρχία της ε, Ρώμης έχει την άποψη και είχε και έχει και σήμερα ότι θα πρέπει ο Επίτροπος ε, αυτός ο έκτακτος να επανεξετάσει αυτή την περιοχή για να δει αν καλύπτονται οι ανάγκες της περιοχής της Ρώμης και κυρίως ε, να μας δώσει περισσότε, πιο περιστατημένες μελέτες και περισσότερα στοιχεία τα οποία θα μας επιτρέπουν να κάνουμε μια πλήρη συνεκτική και ε, διεξοδική αξιολόγηση της περιοχής για να δούμε κατά πόσον μπορεί να δημιουργηθεί αυτή η χωματέρη η οποία θα ήθελα να υπενθυμίσω για να καθησυχάσω και τους αναφέροντες ότι ούτως ή άλλως θα πρόκειται για μία χωματερή προσωρινής φύσεως η αλλως θα προκειται για μια χωματερη προσωρινη φυσεω η οποια ε, θα λαμβάνει απόβλητα τα οποία η νομοθεσία τα καθορίζει ως ειδικά απόβλητα, μη επικίνδυνα και θα είναι αστικά απόβλητα τα οποία θα έχουν τύχει προηγούμενη επεξεργασία και θα έχει γίνει μηχανικό διαχωρισμό και βιολογική επεξεργασία τη οργανική πτυχή των αποβλήτων. Δηλαδή, σε αυτή τη χωματερή, με άλλα λόγια, ούτως ή άλλως δεν θα φτάνει το οργανικό τμήμα των αποβλήτων που είναι το επικίνδυνο τμήμα που δημιουργεί ε, σημαντικά προβλήματα και περιβαλλοντικής αλλά και υγειονομικής φύσεως διότι είναι το τμήμα των αποβλήτων που ε, κατά την υποβάθμισή τους ε, περιλαμβάνουν είτε ε, μολυσματικά στοιχεία που μπορεί να μολύνουν τον, τον υδροφόρο ορίζοντα ή μπορεί να περιέχουν αέρια ε, τα οποία ε, μπορεί να προέρχονται από επικίνδυνες και μολυσματικές ουσίες. Δεν αφορούν όμως αυτά τα απόβλητα. Ε, για να ολοκληρώσουμε όλη αυτή τη συζήτηση για το κατά πόσον είναι κατεπίγουσα η, ε, διαχείριση των αποβλήτων στη Ρώμη, εμείς στη Ρώμη αντιλαμβανόμαστε πλήρως την τον προσανατολισμό του Υπουργού Κλίνη που είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο για τη Ρώμη το οποίο υπέβαλε και στην ε, περιφέρεια της διαχείρισης του Δήμου ε, και ε, στη Ρώμη επιτέλους θα υπάρξει ένα σοβαρό σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων, θα υπάρχει διαχωρισμός των αποβλήτων στην κάθε οικία για να μπορέσουμε να έχουμε υψηλά επίπεδα ε, και διαχείρισης των αποβλήτων ε, όπου θα γίνει το διαχωρισμό στο σπίτι και θα χρησιμοποιούνται και ε, οι χώροι υγειονομικής ταφής ε, των αποβλήτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Ρώμης. Είναι τέσσερις, δύο δημόσιοι και δύο ιδιωτικοί και έτσι θα μπορέσουν να ολοκληρωθεί ικανοποιητικά και σύμφωνα με την νομοθεσία και με πλήρη περιβαλλοντική προστασία το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων στη Ρώμη. Επομένως, εμείς ε, υποστηρίζουμε πλήρως αυτό το σχέδιο το οποίο συνάδει και με τις ε, κατευθυντήριες γραμμές της ε, περιοχής της Ρώμης ε, που ζητά να γίνεται κατοίκον διαχωρισμός των αποβλήτων σε όλη την περιοχή της Ρώμης διότι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή τη μορφή ο διαχωρισμός είναι ο μόνος τρόπος να γίνεται ασφαλός και νομίμως ε, η διαχείριση των αστικών αποβλήπων στη Ρώμη και στην ευρύτερη περιφέρεια. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να ξεκινήσει τώρα η συζήτηση και να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μιλάνα. Ένα λεπτό προσοχή, διότι έχουμε μια κατάσταση Πρόκειται για κάτι βέβαια που αφορά την ευρύτερη αντιπαράθεση στη χώρα, αλλά η Επιτροπή μας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να το τονίσω, βρίσκεται ενώπιον του γεγονότος ότι ε, πρέπει να δράσουμε ή να μην δράσουμε για ένα θέμα. Εγώ δεν θα μπω στην ουσία. Αφενός οι πολίτες έχουν ε, καταθέσει μια αναφορά που λέει ότι υπάρχει μια περιοχή ιστορικής σημασίας, πολιτιστικής σημασίας, ε, είναι πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO χαρακτηρισμένη που μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο. Ο Επίτροπος μας είπε ότι είναι αρκετά μακριά, αλλά τέλος πάντων είναι δυνητικά επικίνδυνο από περιβαλλοντική σκοπιά και μπορεί να ε, υποβαθμιστεί και η αρχαιολογική του αξία. Υπάρχει και ένα ολόκληρο γραφειοκρατικό δε ζήτημα από την άλλη πλευρά. δείτε και τη χώρα έχει να κάνει και με το ποιο πρέπει να κάνει τι. Εγώ άκουσα μια καταγγελία. Οι πολίτες μας λένε στην ουσία ότι χρησιμοποιείται αυτός ο επίτροπος για να αναλάβει μια απόφαση για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε διαδικασίες και δεσμεύσεις που εμείς ουσιαστικά στην Ευρώπη κατά κάποιο τρόπο έχουμε επιβάλει μέσω της οδηγίας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την οδηγία για την προστασία του περιβάλλοντος. Ε, η Επιτροπή μας λέει ότι το μελετάει το ζήτημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι κατεπήγον το ζήτημα και κυρίως θα πρέπει να καταλάβουμε εάν πρέπει εντός εισαγωγικών όχι να ξεκινήσει μια διαδικασία επί παραβάση, αλλά μια διαδικασία στην οποία το καινοτόμο στοιχείο το οποίο επισέρχεται στη συζήτηση είναι η αξιολόγηση μιας πολιτιστικής κληρονομιάς τη UNESCO, δηλαδή μιας περιοχής του οποίου η αρχαιολογική, ιστορική, περιβαλλοντική και καλλιτεχνική αξία είναι αναγνωρισμένη και μάλιστα στην Ιταλία που έχουμε πολλές τέτοιες αντίστοιχες περιοχές, μας ενδιαφέρει εντό εισαγωγικών ε, αυτό περιλαμβάνεται στην αξιολόγηση περιβαλλοντικού αντικτύπου ή όχι. Και θα ήθελα να θέσω αυτό το ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι βρισκόμαστε στα όρια της ερμηνείας ε, του κατά πόσο μπορούμε να δράσουμε εμείς. Αυτή η απάντηση λοιπόν που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που λέει ότι θα μας υποβάλει γραπτός, λαμβάνει υπόψη και την πτυχή αυτή, διότι πέρα από το γεγονό ότι ε, μας είπατε ότι το θέμα αυτό είναι υποέλεγχο έλεγχο, αλλά το είναι υποέλεγχο έλεγχο της ε, ε, των κανόνων μα και το κατά πόσο το τηρεί ένα κράτος ή λαμβάνουμε υπόψη και το θέμα αυτό, διότι το θέμα αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η πρόταση που κάνω εγώ προ την ε, Πρόεδρο και του άλλου συναδέλφου είναι να μην ανοιχτεί αυτή η αναφορά, ώστε η σημερινή ευκαιρία να μας δώσει και την ευκαιρία να εμβαθύνουμε. το γεγονός ότι ο παρόν υπουργό Περιβάλλοντος στην Ιταλία προτείνει και κάτι άλλο και πρέπει να δούμε από εκεί και πέρα τι θα κάνουμε και να είμαστε διατεθειμένοι το θέμα αυτό να το εμβαθύνουμε, ε, να χρησιμοποιήσουμε τη σημερινή ευκαιρία και να προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει το θέμα αυτό το οποίο έχει ε, δημιουργηθεί ως τώρα και ε, έχει ληφθεί υπόψη, να λάβει και δεόντως υπόψη αυτή τη συνιστόσα οι πολίτε λένε ότι πέρα από τις σωσμέ, διότι τα σπίτια μας θα είναι στα 300 μέτρα, αλλά τέλος πάντων αυτό ίσως θα μπορούσε να ε, ρυθμιστεί και από ο τύπο τη χωματερή που μας περιέγραψε ο μηχανικός της περιοχής, να ληφθεί υπόψη και το άλλο γεγονό ότι έχουμε ένα αρχαιολογικό μνημείο αυτή τη σημασία, το οποίο δεν θα πρέπει να το περιβλάπουμε. Θα πρέπει να γίνει με αξιολόγηση και για το θέμα αυτό από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προτείνω λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η απάντησή τη να, να μην είναι η συνήθι γραφειοκρατική απάντηση που θα μα λέει Λάβαμε αυτό, ζητήσαμε αυτό, διότι αυτέ τι απαντήσει παίρνουμε συνήθω. Ε, ετοιμάσαμε έκθεση, κάναμε αυτό, επαληθεύσαμε ότι συνάδει με το τάδε, ξέρω εγώ. Και γίνονται σεβαστοί όλοι αυτοί οι κανόνες και ε, θα πρέπει όμως να υπάρχει και μία αντικειμενική αξιολόγηση για το τι σημαίνει απόβλητο, τι σημαίνει χωματερή ε, σε μία περιοχή που για μένα δεν έχει διαφορά τα 700 μέτρα ή τα 2 χιλιόμετρα, διότι νομίζω ότι οι επιπτώσεις δεν αλλάζουν. Αν περάσουμε από τα 700 μπορεί να υπήρχε διαφορά, αλλά είτε 700 είτε 2 χιλιόμετρα είναι διαφορετικά. Ευχαριστώ κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομα θα πω ότι έχω σοκαριστεί. Βρισκόμουν στην Επιτροπή που πήγε στην καμπάνια και πήραμε το μήνυμα ότι ε, ε θα ανοίξουμε για τα πάντα, φωνάζοντας ακούγαμε ε, για τους διεθνείς κανόνες, τους ευρωπαϊκούς κανόνες, τους ιταλικούς κανόνες. Ε, έκτακτη ανάγκη. Στην Βίλα του Αδριανού πηγαίνοντας εκεί που ε, την είδαμε όλοι μας και στην περιοχή του Βεζουβίου. Ζητώ συγγνώμη. Ε, περιμένετε πραγματικά ότι θα υπάρχει ενδιάμεση φάση και ότι θα καθαρίσει και θα ξαναγίνει πάλι. Πραγματικά θα σταματήσω εδώ, αλλά να πω ότι η Κομισιόν πρέπει να είναι πιο ειλικρινής εδώ και να ζητήσει από την Ιταλία να μην πιστή στην οδηγία. Δεν είναι είτε η καύση είτε χιτά το ερώτημα. Πρέπει να ξεκινήσετε την ανακύκλωση, τη συλλογή, ε, όλες αυτές τις διαδικασίες περιλαμβάνοντας τους πολίτες. Συναντήσαμε εκεί τους πολίτες και πραγματικά έχετε καλούς πολίτες στην Ιταλία αλλά τους βάζετε στην άκρη. ζητώ λοιπόν και από εμά και από την Επιτροπή να είμαστε πολύ πιο αυστηροί εδώ. Αν δεν κάνουμε τίποτα, πραγματικά ε, δεν θα πρέπει ε, να πιστεύουμε ότι η διαδικασία αυτή είναι προσωρινή, θα είναι μόνιμη και θα θάψει την Ιταλία στα σκουπίδια. Ευχαριστώ. Δίνω δύο λεπτά ε, χρόνο για να απαντήσετε. Και μετά ένα λεπτό. Έχετε το λόγο. Ένα λεπτό στον Επίτροπο για να απαντήσει και μετά η αναφέροντος. Ε, να σταθώ μόνο στην τελευταία σας παρέμβαση. Εμείς δεν έχουμε καμία πρόταση να σας πω ότι εγώ είμαι από την Νάπολη καταρχάς. Ε, είδα τι έγινε στην Νάπολη και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε η Ρώμη να γίνει σαν την Νάπολη. Ε, και λυπάμαι ήθελα να σας διαβεβαιώσω ε, και προς αυτή την κατεύθυνση, ότι δεν θα γίνουμε Νάπολη. Κρίμα που σηκώνεστε από τη θέση σας και δεν ακούτε την απάντηση. Δεν, μπορούμε να, δεν μπορώ να είμαι σε δύο μέρες την ίδια ε, στιγμή και αλλάξατε την ημερήσια διάταξη. Τι να κάνω, λέει η κυρία Άουκεν εκτό μικροφώνου. Γεια σα. Θα έρθω μετά και θα μου πείτε τι έγινε. Comunque non sono qui per fare Τέλο πάντων, εγώ δεν ήρθα εδώ για να ξεκινήσω διαμάχε, ε, διότι δεν έχω καμία πρόθεση να ξεκινήσει και διαμάχη ε, σε προσωπικό επίπεδο. Η πρόθεση της Ιταλικής κυβέρνησης και κυρίως η δική μου και των αρχών της Ρώμης είναι να ολοκληρωθεί αυτή η έκτακτη κατάσταση το συντομότερο δυνατόν. Εμείς σας ζητάμε λίγο χρόνο, 1,5-2 χρόνια, για να μπορέσουμε από εκεί και πέρα να περάσουμε σε αυτό που έλεγε ο κύριος Μιλάνα και η κυρία Άουκεν, να περάσουμε στην ανακύκλωση σε ένα σχέδιο το οποίο ούτως ή άλλως έχει παρουσιάσει ήδη η περιφέρεια της Ρώμης. Ζητάμε λίγο χρόνο για να το θέσουμε σε εφαρμογή. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος τώρα στους ε, δύο αναφέροντες. Ένα λεπτό καθένας, ε. Πολύ σύντομο δεν θέλω να ξεκινήσω στοιχείες για ε, συζητήσεις για δεδομένα και το καθεξής, αλλά το ξέρουν όλοι ότι η βιολογική μηχανική επεξεργασία των αποβλήτων αυτή τη στιγμή δεν επαρκεί για να ικανοποιήσει ε, σε σύντομο χρονικό διάστημα την ε, διαχείριση των επεξεργασμένων αποβλήτων. Και υπάρχει και μια ανομαλία η οποία σχετίζεται από την έλλειψη εμπειρίας, όπως είπε και ο, ο κύριος της νομαρχίας, που δεν φταίει αυτός, αλλά είναι δεδομένο. Το άρθρο 2, στο παράγραφο 4 της ε, νομοθεσίας, λέει ότι ο αρμόδιος επίτροπος αναλαμβάνει τα θέματα της διαχείρισης ε, για τους χώρους επεξεργασίας και τη διάθεση των αποβλήτων στην περιοχή που καθορίζεται και θα πρέπει όλα αυτά να γίνονται σε συγκεκριμένα χρονικά διάστημα εντός 30 ημερών και ε, υιοθετεί τις απαραίτητες διατάξεις ε, και μέχρι τώρα δεν έχουμε ε, διαπιστώσει ότι έχει ληφθεί κάποια απόφαση και αυτή η ε, απόφαση είναι από το Σεπτέμβριο και αναφερόμαστε μόνο στα απόβλητα αυτή τη στιγμή. Ναι, και εγώ πολύ σύντομα υπάρχει ένας παράγοντας ο οποίος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η τελευταία παράταση για τη χωματερή της Μαλαγκρότα τελειώνει τον Ιούνιο. αυτή τη στιγμή δεν γίνεται να γίνει πλήρης διαχείριση των αποβλήτων βάσει των σχεδίων. Υπάρχει ανάγκη να μην υπάρχουν ε, επεξεργασμένα, μη επεξεργασμένα απόβλητα, ε, διότι πρέπει να γίνεται, το ζητά και η Ευρώπη και υπάρχουν και συγκεκριμένε ε, ζημίες. Και υπό αυτό το πρίσμα πώς είναι δυνατόν να μας λέτε ότι έχουμε προσωρινή χωματερή αυτού του είδους. Αυτά, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι απόλυτη σαφή η πρόθεση της Επιτροπής μας. Θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε την αναφορά αυτή. Θέλετε το λόγο? Είχε ολοκληρωθεί η παρέμβαση. Είχαμε ολοκληρώσει, αλλά τέλος πάντων. Ευχαριστώ. Δυστυχώς ε, ταυτόχρονα είχαμε και ε, μία συνάντηση με τους ε, Ευρωπαίους υπεργούς και εγώ ως αρμόδιος ηγητής δεν μπορούσα να λείψω, την είχαμε οργανώσει, θέλαμε να πάμε και όλοι, λέει ο κύριος Μιλάνα. Πρόκειται για ένα στοιχείο το οποίο δεν συζητήθηκε και θα ήθελα να το πούμε εδώ. Εγώ είχα γράψει στο νομάρχη τότε και είχα ζητήσει πληροφορίες για την ιδιοκτησία των χώρων τους οποίους συζητάμε εδώ στην Ακρόαση. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και πρέπει να πω στον Ομάρχη ότι σε εκείνη την επιστολή η οποία ε, έχει αποσταλεί πριν από αρκετού μήνες δεν έλαβα καμία απάντηση. Και ε, νομίζω ότι αυτό δεν είναι σωστό και για τις ε, διοργανικές σχέσεις που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ ενός εκπροσώπου των, ε, ε της τοπικής και ενό ευρωβουλευτή, αλλά και γιατί λείπει ένα στοιχείο από τη συζήτηση το οποίο νομίζω ότι έχει και μια κάποια βαρύτητα. Ο νομάρχης. ο Επίτροπος. Δεν θυμάμαι εγώ την επιστολή σας, αλλά απάντησα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, και στη Γερουσία και όπως απάντησα και σε αυτού θα μπορούσα να απαντήσω και σε εσά. Δεν είχα λόγο να μην του απαντήσω. Άρα θα σας απαντήσω. Αν μου ξαναστείλετε την επιστολή σας, εγώ θα φροντίσω να λάβετε την απάντηση. Ε, λοιπόν, έχουμε μια άτυπη ανταλλαγή μεταξύ του συναδέλφου και του επιτρόπου και να σας πω ότι Ίσως θα έπρεπε όλα τα ε, έγγραφα τα οποία θα πρέπει να περιληφθούν για τη συζήτηση θα πρέπει να τα αποστείλετε και στην Πρόεδρο για να τα δώσει από εκεί και πέρα στα μέλη τα οποία θα πρέπει να λάβουν απόφαση. Έλεγα προηγουμένως λοιπόν ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα όσα ζητούν τα μέλη της Επιτροπής είναι να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Υπάρχουν κάποιες ασάφειες και αβεβαιότητες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ήδη ότι θα επαληθεύσει και ε, κατά πόσον είναι νόμιμη η διαδικασία της αξιολόγησης αντικτύπου ε, για να εντοπιστούν ποιες θα είναι οι περιοχές όπου θα δημιουργηθούν χιτά και αυτός επίσης και τι γίνεται με την διαβούλευση και την ακρόαση των πολιτών όταν έχουμε πρωτοβουλίες οι οποίες είναι παρεμβατικής φύσεως και για το περιβάλλον αλλά και για την κοινωνική ζωή των πολιτών και ελπίζουμε να μπορέσουμε να λάβουμε την απόφαση η οποία μας είπατε ότι θα ε, μας αποσταλεί και ελπίζουμε η σημερινή συζήτηση να έδωσε και επιπλέον στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα οποία θα μπορούσε να εντάξει στο έγγραφο το οποίο θα μας διαβιβάσει και φυσικά και στη... θα βοηθήσει και την Επιτροπή μας να κάνει την αξιολόγησή της. Να ενημερώσω εδώ τους εκπροσώπους ε, των δύο οργανώσεων που κατέθεσαν την αναφορά ότι εμείς ε, σκοπεύουμε τον Οκτώβριο νομίζω να κάνουμε μια επίσκεψη στην Ιταλία και ε, μεταξύ άλλων θέλαμε να αποφασίσουμε ε, και να πάμε να δούμε και τι γίνεται σε αυτά τα οποία, ε, στην περιοχή στην οποία μας είπατε και να δούμε αν όντως ισχύουν όλα αυτά. Δεν θα πάρουμε βέβαια ε, μέτρο για να μετρήσουμε την απόσταση των 2.700 μέτρων, αλλά θα εκμεταλλευτούμε αυτή την επίσκεψή μας για να δούμε πόσο δύσκολη είναι αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ τις αρμόδιες τοπικές αρχές που ήταν παρούσες, ευχαριστούμε και τους πολίτες που μας υπέβαλαν αυτή την αναφορά και μας έδειξαν τι δυσκολία υπάρχει για πολλωστή φορά στην Ιταλία και ολοκληρώνεται το σημείο αυτό προς το παρόν. Έχουμε ήδη καθυστερήσει αρκετά λεπτά τη συνεδρίαση. Γι' αυτό λοιπόν σας προσκαλώ να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Προστασία και την ε, Ευζοία των Ζωών 2012-2015. Ε, ο κύριος ε, Βοστινάρου είναι ο εισηγητής. Θέλετε το λόγο? Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, το είπα ήδη κατά τη διάρκεια της, ε, του σχεδίου της γνωμοδότησης στην Επιτροπή Γεωργίας ε, για το θέμα της υγείας και της ευζοίας των ζώων. Ε, προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε με τους ε, πολίτες ε, για αυτές τις ε, τέσσερις αναφορές που έχουμε συζητήσει εδώ. Έχουμε ακόμα τις δραματικές εικόνες στο, μπροστά στα μάτια μας. Προσπάθησα όλες οι αναφορές να είναι ισόρροπα, να προσιαστούν ισόρροπα και επίσης να είμαι δίκαιος ω προς τα συμφέροντα που εκπροσωπούνται σε αυτό το θέμα. Να πω λοιπόν ότι δεν υπάρχει κοινοτική νομοθεσία ειδικότερα για την προστασία και την ε, υγεία των ζώων, ε, ειδικότερα για τα ε, αδέσποτα και για τα ε, οικόσιτα ζώα. όλο και πιο συχνά λοιπόν τα θέματα αυτά ε, έρχονται ε, στην Επιτροπή Αναφορών. Θα ήθελα λοιπόν ε, να ζητήσουμε να υπάρχουν τα ελάχιστα στάνταρ για την προστασία των ζώων κατά τις μεταφορές μέσα στα πλαίσια μιας νομοθετικής διαδικασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα η Επιτροπή μας ανέβαλε μία έστειλε μία ψηφοφορία στην, στην Ολομέλη. Αυτό δείχνει πραγματικά πόσο είμαστε σε αυτό το θέμα ε, ταγμένοι. Σήμερα ελπίζω να μπορέσουμε να ψηφίσουμε αυτό που είναι σημαντικό για τους πολίτες. Θα πρέπει να υπάρχει ε, αυστηρή νομοθεσία σχετικά με, τις τα επιστημονικά πειράματα στα ζώα, για παράδειγμα. Στο μέλλον σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Ευχαριστώ όλους τους εκπροσώπους της κοινωνίας των ε, πολιτών που έδειξαν την ευαισθησία τους σε αυτό το θέμα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφε. Μιλήσατε για τους πολίτες. Θα ήθελα τώρα να ξεκινήσει η ε, ψηφοφορία. Ε, τροπολογία 1 από τον συνάδελφους Τέιλορ, Ραούλ Ρουέντα, υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται τροπολογία 3, παράγραφος 1, υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 2 Παράγραφος 1α, Τέιλορ, Ραούλ, Ρουέντα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ζητώ συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος. Ε, αρχίζει η ψηφοφορία για την τροπολογία 2 παραγραφός 1 και Κέιθολ, Ραούλ και Ρωμέρα και Δρουέδα. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Μάλλον υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Sì. Allora, proviamo. Funziona? Okay. Avete votato Ψηφίσανε όλοι, κλείνει η ψηφοφορία. Δεν έχει κλείσει η ψηφοφορία. Θα προσθέσουμε και την ψήφο του συναδέλφου Ιντορκάης. Δεν λειτουργεί. Ψήφισαν 15, ε, υπέρ 5, 9 κατά, απορρίπτεται και ο κύριος Ιτουργκάης που είναι κατά 10 λοιπόν κατά, άρα απορρίπτεται η τροπολογία. Τροπολογία 6 παραγραφός 2, Βέρτμαν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4, Τέιλορ και Ραούλ Ρέδα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5 παραγραφός 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 7, παράγραφος 2α, ε, φάξας υπέρ, κατά, αποχές, απαρρίπτεται. Παράγραφος 3, 9, τουργκάες, έχει κάνει μια προφορική ε, τροπολογία. Υπάρχει κάποιος που να είναι κατά στην τρο... της προφορικής τροπολογίας. Όχι. Ωραία. Ψηφίσουμε την τροπολογία 9, όπως έχει ε, αλλαχθεί υπέρ κατά αποχές. Ας κάνουμε τον έλεγχο. Θέτουμε σε ψηφοφορία την 9 του συναδέλφου Ιτουργκάης. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 17 ψήφισαν 11 ε, ε, υπέρ, ε, άρα εγκρίνεται. 8 παραγραφός 3, συνάδελφος. Επειδή λοιπόν έχουμε δεχτεί αυτήν, πάμε στη 10 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται τροπολογία 11, παραγραφός 4, οι ίδιοι συνάδελφοι υπέρ, κατά, Δεν έχετε πια μετάφραση. Το μικρόφωνο. Δεν σας ακούμε. Ζητείτε να γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση. Μάλλον δεν υπήρχε ε, η μετάφραση σε κάποια γλώσσα. Στα αγγλικά. Μπορούμε να ξαναψηφίσουμε. Πάμε πίσω στην τροπολογία 10 λοιπόν, η 8 καταπίπτει. Ηλεκτρονική. Άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 2 υπέρ, 15 κατά. Τροπολογία 11, παράγραφος 4. Τέιλος, Σόκεν, Περ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12, παράγραφος 4α, Πάκτσας, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14, παράγραφος 5, υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 13 παράγραφος 5 Βαλέσα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 παράγραφος 5α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 Τερλόρο Ρόκεν Ραούλ Ροέδα παράγραφος 6 χωριστή ψηφοφορία πρώτο μέρος υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 17 παράγραφος 7, φως Γιάρ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 18 παράγραφος 8, Τέιλορ Ραούλο Ροέδα, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Ok, verifichiamo il paragrafo, l'emendamento 18. Επιβεβαιώνουμε την 18 παράγραφος 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. 2 υπέρ, 15 κατά. Απορρίπτεται. Με την επαλήθευση είμαστε πιο ήσυχοι. Τροπολογία 19 για παράγραφος 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 έχει αποσυρθεί, 24 παράγραφος 10 βαλεάν υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 21, παράγραφος 10, Βαλέσα υπέρ. Ε, καταπίπτει. Όχι, μόνο αν εγκριθεί η άλλη. Εντάξει. Τροπολογία 21, Βαλέσα, παράγραφος 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22, για παράγραφος 10, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23, Τέιλο Ρόκεν Ροέδα, παράγραφος 10, σε χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Τροπολογία 25, Taylor Oaken Ρουμέδα, 11α, υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 26, Taylor Oaken Ρουέδα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27, Γιάρ, παράγραφος 13, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται να κάνουμε έναν έλεγχο για την τροπολογία 27, παράγραφος 13, άρχεται η ψηφοφορία. Δεν άρχισε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Δώδεκα υπέρ εξκατά εγκρίνεται. Τροπολογία 28, παράγραφος 13. Όχι. Επειδή εγκρίναμε την προηγούμενη τροπολογία κατά πάμε στην 29 Taylor Rock και Veruenda, παράγραφος 14 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 30, παράγραφος 14 Βάλεν, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31, Τέιλο με Ρομεβερουέδα 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε όλο το έγγραφο. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. 17 υπέρ ένα κατά κλείνεται. Κλείνει η ψηφοφορία. 17 υπέρ, καθένα κατά, κλείνει η ψηφοφορία. you Κύριε Ο κύριος Μπουσούτιλ ζητά λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα απλώ να καλωσορίσω μία ομάδα ε, επισκεπτών που έχουν έρθει από την περιοχή μου στη Μάλτα. Του ευχαριστώ πολύ για την παρουσία του εδώ. Πολύ ευχαριστώ και εμεί ε, καλωσορίζουμε την αντιπροσωπεία που έχει έρθει εδώ από τη Μάλτα. Ελπίζουμε να του ευχαρίστησαν οι εργασίες μας. Reluăm ședința. Vă rog frumos, trecem în continuare la subiectul următor, petiția numărul 1675 din 2. Θα τώρα στην αναφορά 675-8 από τους πράσινους της Βουλγαρίας σχετικά με τη λεγόμενη διαδικασία ανταλλαγής γεών και τη διαφθορά στη Βουλγαρία. Δεν είναι ο αναφέρον παρόν, θα εκπροσωπηθεί όμως από εκπροσώπους του Υπουργείου Γεωργίας της Βουλγαρίας, την κυρία Νικολόβα, τον κύριο Ιώσιπόβ και τον κύριο Τσουμιρτζέμ. Κυρίες και κύριοι, έχετε το λόγο με τη σειρά που επιθυμείτε εσείς. Din partea Ministerului Agriculturii, aveți... Λοιπόν, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας της Βουλγαρίας έχουν τον λόγο. The petitioners are not present, I already said. ο δεν είναι εκείνος που θέλετε να φορά, δεν είναι παρόν. Το κατέστησα σαφές νομίζω. Κατέστησα απόλυτα σαφές ότι το άτομο που κατέστησε την αναφορά δεν είναι παρόν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 ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας θα ήθελα να λάβω το λόγο για αυτή την αναφορά. Έχει σχέση με μια πρακτική που αφορά τις ανταλλαγές εκτάσεων. Είναι μια πρακτική η οποία από τον, το 2003 στο 2009 ήταν αρκετά συχνή. Μετά από την υποβολή της αναφοράς απαγορεύθηκε αυτή η πρακτική. Και υιοθετήθηκε αυτή η απόφαση από το σημερινό ε, κοινοβούλιο και δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Βουλγαρίας. Ποια είναι τώρα η θέση της κυβέρνησης. Όσον αφορά λοιπόν αυτή την ανταλλαγή γεών, εκτάσεων, κανένα από τα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 37 για ε, τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεν ισχύει. Η Βουλγαρία αποτελεί αντικείμενο μιας επίσημης έρευνας την οποία διεξήγαγε η Επιτροπή το 2011 μια έρευνα για τις ε, ενισχύσεις, ε, δημόσιες ενισχύσεις που ε, υπήρχε υπόνοια ότι υπήρχαν στην περίπτωση των ανταλλαγών εκτάσεων. Επτά ημέρες μετά από την εκλογή της κυβέρνησης, ο Υπουργός Γεωργίας, ο κ. Σμιτνόφ, έδωσε εντολή απαγόρευσης προσφυγής όσον αφορά την ανταλλαγή εκτάσεων και επίσης το Κοινοβούλιο υιοθέτησε μια απόφαση όσον αφορά την αναστολή της αλλαγής χρήσης γης για εκτάσεις που ανήκουν στο κράτος. το Μάρτιο του 2011 έγιναν ε, ε, διαβουλεύσεις με οργανισμούς του περιβάλλοντος το άρθρο 35 του νόμου απαγορεύει πλήρως την ανταλλαγή εκτάσεων α, για δασικές εκτάσεις. Ε, τι Και επίσης απαγορεύεται η αλλαγή στη χρήση γης. θεσπίστηκε και άλλη νομοθεσία εφαρμοστική της πρώτης που ορίζει, που αναφέρεται στις εκτάσεις που υπήρξαν αντικείμενο ανταλλαγή. Και στην εγγραφή αυτών των, των εκτάσεων που έχουν ανταλλαγή στο κτηματολόγιο. Νομίζω λοιπόν ότι η Βουλγαρία ανταποκρίθηκε σε αυτό το αίτημα στα πλαίσια ε, του μηχανισμού συνεργασίας και επαλήθευσης επόμενη τις δεσμεύσεις της που προκύπτουν από το 2011. Όσον αφορά λοιπόν ε, τις ανταλλαγές εκτάσεων, ε, αυτές αφορούν μεταξύ 5 και 9.000 εκτάρια. πρέπει να εξηγήσουμε ότι μεταξύ 2003 και 2009 οι ανταλλαγές εκτάσεων ανήλθαν συνολικά σε 3,3 εκτάρια μετά την προσχώρηση της Βουλγαρίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η ποσότητα έφτασε το 2.400. Ως αποτέλεσμα, η χώρα έλαβε περίπου 14 εκατομμύρια λεβ Βουλγαρίας ως, ε, αποτέλεσμα της μείωσης των ανταλλαγών εκτάσεων. Στην πράξη όμως, η αλλαγή χρήσης γης, δηλαδή από δασικές εκτάσεις σε μη δασικές, άρχισε να ισχύει από τον Ιανουάριο του 2009. και αφορά 460 εκτάρια. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι αποφάσισε το Εθνικό Κοινοβούλιο η απόφαση μάλλον αυτή έχει γίνει πλέον νόμος του κράτους και σχετικά με την αναφορά ε, στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βουλγαρίας και σύμφωνα με την απόφαση αυτού του δικαστηρίου η βουλγαρική κυβέρνηση αποφάσισε να απαγορεύσει εντελώς τις ανταλλαγές δασικών εκτάσεων Καταλήγοντας, θέλω να σας πω το ύψος των απολειών που, ε, στις οποίες αναφέρεται ο αναφορά ανέρχεται σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά αυτό το ποσό είναι υπερβολικό. Έχει υπερβάλλει. δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η θέση της Δημοκρατίας Βουλγαρίας και ιδιαίτερα του Υπουργείου Γεωργίας είναι η εξής όλες οι ανταλλαγές για την περίοδο 2003-2009 έχουν ελεγχθεί λεπτομερέστατα από μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων ad hoc και αυτή τη στιγμή ε, συνεχίζεται αυτή η έρευνα για τις ανταλλαγές εκτάσεων πράγμα το οποίο επαληθεύεται από το ανώτατο δικαστήριο από τον, της ε, Βουλγαρικής Δημοκρατίας έχουν γίνει 25 ε, αρχικοί έλεγχοι με βάση το υλικό που έχει παράσχει το Υπουργείο Γεωργίας. Υπάρχουν και διαφορές, αλλά ακόμα δεν ε, ε, υπάρχει καμία καταδίκη. Ευχαριστώ. Τώρα δίνω το λόγο στους άλλους εκπροσώπους του Υπουργείου ε, Γεωργίας Βουλγαρίας τη σειρά που εσείς επιθυμείτε. No, no. Da, deoarece niciunul dintre dumneavoastră nu dorește să mai ia cuvântul, dau în continuare cuvântul Comisiei Europene să ne prezinte από ό,τι κατάλαβα, δεν θέλετε να μιλήσετε. Δίνω το λόγο λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα μα παρουσιάσει την άποψη της Επιτροπής. Έχετε το λόγο, κύριε μου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως αναφέρθηκε ήδη από τον εκπρόσωπο τη Δημοκρατία Βουλγαρίας, έχει ανοίξει μια διαδικασία διερεύνηση αυτής της κατάσταση όσον αφορά τις ε, ανταλλαγές δασικών εκτάσεων. Αυτό δεν αφορά με μονομένες ανταλλαγές εκτάσεων, αλλά η Επιτροπή ε, προσπαθεί να διερευνήσει το σύστημα, το διοικητικό σύστημα, προτού σταματήσουν να απαγορευτούν οι ανταλλαγές εκτάσεων. Αυτή η μέθοδος, δηλαδή οι, οι τιμές ε, που αφορούσαν τις ε, ανταλλαγές εκτάσεις, δεν είχαν οριστεί αρχικά σύμφωνα, ας πούμε, με εκείνο το οποίο θα λέγαμε ε, τις τιμές, τις αγορές τιμές, αλλά είχαν βασιστεί σε μια διοικητική μέθοδο. Αυτή τη στιγμή η Επιτροπή διερευνά κατά πόσον αυτή η διοικητική μέθοδος καθορισμού των τιμών ή μάλλον οι παρατυπίες και η έλλειψη ορισμένων συντελεστών που είχαν χρησιμοποιηθεί καταλήγει σε τιμές που δεν ε, βρίσκονται κοντά στις αγορές τιμές. Αν αυτό συμβαίνει, τότε πιθανόν να υπήρξε ένα ε, ε, οικονομικό πλεονέκτημα το οποίο δεν έπρεπε να υπάρχει και, το, και τελικά θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ότι αυτές ήταν κρατικές ενισχύσεις. Σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο των συνθήκων. Στα πλαίσια αυτής της ε, επίσημης διαδικασίας έρευνας, αυτό δεν προδικάζει, εν πάση περιπτώσει, τη θέση της Επιτροπής. Αλλά δίνει την δυνατότητα σε τρίτα μέρη που ενδιαφέρονται να δώσουν τα σχόλιά τους επάνω στα θέματα που αναλύει η Επιτροπή. Σε αυτή την περίπτωση της ανταλλαγή συνταξιτικών εκτάσεων λάβαμε πολλά σχόλια από 25 ενδιαφερόμενα μέρη που αναλύονται τώρα από την Επιτροπή. Με βάση αυτά τα σχόλια και φυσικά με βάση τα σχόλια της Βουλγαρίας η οποία έχει τη δυνατότητα να σχολιάσει την απόφαση και τα σχόλια που έχουν σταλεί από τρίτα μέρη, η Επιτροπή δική μας ε, θα εξετάσει τα σχόλια και θα χρησιμοποιήσει αυτά και άλλα στοιχεία για να καταλήξει κατά πόσον αυτό συνιστά ε, κρατικές ενισχύσεις εάν αποφασίσει η Επιτροπή ότι πρόκειται για κρατικέ ενισχύσει λόγω τη διοικητική τιμή που ορίζεται και λόγω ε, τη μη χρήση των συντελεστών, η Επιτροπή θα αποφασίσει κατά πόσον αυτέ οι κρατικέ ενισχύσει συμβαδίζουν ή είναι συμβατέ με την εσωτερική αγορά. Εάν τελικά αποφασίσουμε ότι αυτέ οι κρατικέ ενισχύσει δεν είναι συμβατέ, τότε η Δημοκρατία τη Βουλγαρία θα κληθεί ε, να επιστρέψει τι κρατικέ ενισχύσει που ελήφθησαν. Συνεπώς, είναι σημαντικό να πούμε ότι εδώ υπήρξαν ορισμένες παρεξηγήσεις. Δηλαδή, σύμφωνα με τη διαδικασία των κρατικών ενισχύσεων, Δεν είναι δυνατόν να επιβάλλει κανείς ε, κυρώσεις σε αυτά τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα κονδύλια δύο κρατικέ Απλώς θα ζητήσει η Επιτροπή να επιστραφούν αυτά τα χρήματα. Όπως είπα όμω, λάβαμε πολλά σχόλια από πολλές τρίτες πηγές και αυτή τη στιγμή αναλύουμε όλες τις πληροφορίες που εστάλησαν σε εμά και στο παρόν στάδιο η Επιτροπή δεν είναι ακόμα σε θέση να καταλήξει για ε, το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας που γίνεται για το κατά πόσον πρόκειται για κρατικές ενισχύσεις. Ευχαριστούμε την εκπρόσωπο της Επιτροπής. Θα ήθελα τώρα να στραφώ στους συναδέλφους. Υπάρχει κάποιος που θέλει να πάρει το λόγο. Θα ήθελα να ρωτήσω στους εκπροσώπους και της Επιτροπής και των βουλγαρικών αρχών εάν αναμένουν μια κατάσταση που είναι πανεμιότυπη, ε, όπου αγόραζαν δασικές εκτάσεις τα άτομα, ε, πληρώντας μόνο 2 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ίσως είναι η φθηνότερη γη στον κόσμο. Αλλά έχετε εκτιμήσει και αυτή την κατάσταση. Διότι στην περίπτωση Μπάνια είχαμε ε, επισκεφθεί αυτό το θέρετρο το οποίο ε, επηρέαζε και τον, ε, την περιοχή Natura 2000 αλλά ήταν μια δραματική, τραγική παρέμβαση, επέμβαση στο περιβάλλον Natura 2000 επειδή είχαν κόψει τα δέντρα, δεν ήταν θέρετρο, με συγχωρείτε, ήταν σταθμός στενοδρομικός. Έκοβαν πάρα πολλά δέντρα για να φτιάξουν καθόδους για σκι και ε, πέρσι ε, εξετάσαμε τη μελέτη που έγινε τόπο από τη Βουλγαρία και η συνάδελφός μου και η Άλκον είχε ε, απαντήσει, αλλά ακόμα οι βουλγαρικές αρχές δεν έχουν απαντήσει γιατί αυτό το θέμα παραπέμπεται σε ελληνικές καλένδες. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να μιλήσει. Αν όχι, δίνω το λόγο στις βουλγαρικές αρχές αν επιθυμούν να προσθέσουν κάτι. Ε, в случая ние вече подчертахме, че всички случаи от 2003 година до 2009 година. Και εμεί αναφέραμε ότι στην περίοδο 2003-2009 όλες οι ανταλλαγές είναι ανταλλαγές δασικών εκτάσεων. με ε, ε, ιδιωτικέ εκτάσεις. Και όλα αυτά έχουν παραπεμφθεί στο ανώτατο δικαστήριο. Λοιπόν, όταν υπάρχει παραβίαση του ποινικού κώδικα, το Υπουργείο Γεωργίας τότε ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές. Όπως είπε εκπρόσωπος Επιτροπής, η έρευνα καλύπτει τα θέματα παραβίαση των συνθήκων του άρθρου 107 διότι παράνομα ε, δόθηκαν κρατικές ενισχύσεις. Μετά από την 1η Ιανουαρίου 2007, όταν γίναμε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Βουλγαρία δεν εφήρμοσε από τότε ε, ε, τον κανόνα των κρατικών ενισχύσεων. Αυτό το αναφέραμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ε, το χρονοδιάγραμμα που αρχίζει από την εποχή που ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μιλάμε για ανταλλαγή δασικών εκτάσεων. Και όλα τα έγγραφα που αφορούν την διοικητική εκτίμηση σύμφωνα με τους κανόνες του 2003 έχουν ε, κατατεθεί στην εισαγγελία και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το θέμα λοιπόν δεν το αφήσαμε κατά μέρο, αλλά διερευνάται από τις ε, βουλγαρικές αρχές και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε σχέση πάντοτε με τις κρατικές ενισχύσεις. Τώρα, η αντιπροσωπεία τη διαφθοράς και του νεποτισμού ε, δεν έχει ακόμα απαντήσει, γι' αυτό συνιστώ να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Δεν έχουμε απαντήσεις. Ερχόμαστε τώρα στην έκθεση της ε, Επιτροπής Πέτσα στο Βερολίνο. Ο κύριος Μάρεξ Σταβίνοφ και ο κύριος Γιώργη Γκάτος είναι παρόντες εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και έχουν το λόγο.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 Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα σας εξηγήσω το περιεχόμενο της αντιπροσωμίας μας, όμως ε, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι εδώ βρισκόμαστε μόνο τρία άτομα από αυτή την αντιπροσωπεία. Και δεν ξέρω αν είναι και πολύ σωστό να συζητήσουμε σήμερα αυτό το θέμα και την ε, αποστολή στο Βερολίνο. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν ποια είναι η γνώμη και των συναδέλφων που είναι μέμλη αυτή τη επιτροπή, αυτή τη αντιπροσωπείας μάλλον. Θέλετε να συνεχίσουμε? ich möchte eingangs noch einmal betonen. Να τονίσω για άλλη μια φορά ότι πραγματικά ευχαριστώ πολύ, ειδικότερα τον κύριο Ότοβα και την ομάδα που προετοίμασε αυτό το θέμα, ακόμα και αν είχαμε άλλη άποψη για κάποια θέματα, θεωρώ ότι τώρα τα πράγματα ε, πήγαν πολύ, κατά και πολύ καλά. Η διαδικασία πήγε καλά και σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω κάποιες προσωπικές παρατηρήσεις και κάποιες ε, ερωτήσεις, αν έχουμε επίσης τη δυνατότητα να ε, καταθέσω δύο τροπολογίες. Η μία έχει να κάνει με το θέμα των ούτως αποκαλούμενων recommendations συστάσεων και που είναι σε συνδυασμό με τα conclusions, συμπεράσματα. Θα ήθελα να μπουν αυτά στη διαδικασία των τροπολογιών, να ενταχθούν, διότι θεωρώ ότι τα συμπεράσματα έχουν μια αξία και είναι και μια πολιτική δήλωση, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ καλό και πρέπει να ενταχθεί στη διαδικασία. Äh, Θεωρώ ότι εγώ προσωπικά ε, δεν μπορώ να καταλάβω πολύ καλά το τελευταίο κομμάτι πριν στα συμπεράσματα που λέει ότι τα μέλη της, αντιπροσωπείας δεν είχαν κάποια ξεκάθαρη εικόνα για το περιεχόμενο των πληροφοριών που πήραν στο Βερολίνο και δεν ήταν και ξεκάθαρες οι αρμοδιότητες. Αυτό δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Αν είναι νόμιμο πραγματικά να, κάνουμε τέτοια, να βγάζουμε τέτοια συμπεράσματα, τότε έχει κάποιο νόημα να μπει στις τροπολογίες. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια διαδικασία ε, πολύ στοχοθετημένη και γι' αυτό σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Συζητήσαμε το θέμα της έκθεσης και ένα πολύ σημαντικό πράγμα αυτή τη στιγμή είναι να έχουμε μια συνένεση παρά τις διαφορές απόψεων. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να επιληθούν μέσα σε μία εβδομάδα και γι' αυτό ε, αναβάλαμε λιγάκι την τελική επιτροπή μέχρι να φτάσουμε σε μία ε, συνένεση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Συνεχίζουμε με τον ε, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έκθεση και το σχέδιο. Μάλλον δεν υπάρχει εκπρόσωπος της Κομισιόν που να θέλει να μιλήσει για το θέμα ή όχι. Ζητώ συγγνώμη. Ναι. Για λόγους διευκρίνησης να πω ότι είναι η πρώτη φορά που ακούω ότι η Κομισιόν ε, εμπλέκεται σε αυτό το θέμα. Δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Η Κομισιόν έχει πάντοτε εδώ εκπροσώπους, ενδιαφέρονται για τη δουλειά που κάνουμε. Δεν αλλάζουν την έκθεση, απλώς παρακολουθούν τη συζήτησή σας. Αυτός είναι ο ρόλος της Κομισιόν σε αυτή την περίπτωση. Uh, I don't think they have αλλά δεν έχουν σκοπό να παρέμβουν στη συζήτηση ούτως ή άλλως από ό,τι φαίνεται. Εκ των προτέρων λοιπόν να σας πω ότι υπήρξε ε, ένα ταξίδι της αντιπροσωπείας στη Ρουμανία, οποία ε, είχε προσκληθεί η Επιτροπή. Ίσως λοιπόν αυτό να μην σας ε, εκπλήσει. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήταν μάλλον δική μου η παρανόηση, γιατί είχα την εντύπωση ότι ε, λέγατε πως ε, η Επιτροπή είχε κάποια θέση ως προς αυτό το ευαίσθητο θέμα και ως τώρα δεν έχει εμπλακεί καθόλου στην διαδικασία. Μάλλον κάπου στο μέλσο είναι το λάθος. Τώρα, σχετικά με την αποστολή στο Βερολίνο, θα πρέπει να αποφασίσουμε ε, για τη διαδικασία που θα ακολουθεί στο εξή. Ε, λυπάμαι που υπάρχουν τόσο λίγα μέλη, που υπάρχουν τόσο λίγα μέλη της Επιτροπής εδώ. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Και πραγματικά θα το συζητήσουμε τόσο λίγοι. Ευρωβουλευτές. Ενημερωθήκαμε ότι αυτό το θέμα δεν θα είναι στην ημερήσια διάταξη σήμερα και αυτό είναι λάθος. Ίσως γι' αυτό δεν είναι εδώ ο κόσμος. Αυτή η αντιπροσωπεία για την προστασία των παιδιών και νεαρών έγινε η αποστολή δηλαδή πριν από έξι μήνες. Έχει να κάνει με τα δικαιώματα των γονέων, ένα ευαίσθητο θέμα. Θέλανε στην ουσία να δουν γιατί υπήρχαν τόσες πολλές αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ειδικότερα δεδομένου ότι υπήρξε και στο παρελθόν μια τέτοια αποστολή. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων και στη συνέχεια αυτών, να επαναλάβω για άλλη μια φορά, η αποστολή δεν είχε ως σκοπό ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν θέλαμε να ε, παρέμβουμε με, στην ε, γερμανική νομοθεσία ή να πάρουμε το μέρος κάποιου. Θέλαμε να δούμε γιατί ε, παραπονούνται οι Ευρωπαίοι πολίτες για αυτήν την υπηρεσία. Και να βρούμε μια λύση. Μιλώ υπό την Αρμοδιότητα μου ως ε, βουλευτής ε, της Επιτροπής ε, Αναφορών. Υπάρχουν διάφορες απόψεις μέσα στην Επιτροπή μας. Ο κ. Μπέκερ είπε ότι δεν είχαμε πάντοτε συμφωνήσει και δεν είχαμε πάντοτε συνένεση. Όταν μιλάμε για συστηματικές παραβιάσεις, δεν σημαίνει ότι όλοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους σε μια υπηρεσία, απλώς υπάρχουν πολλά προβλήματα στη συγκεκριμένη υπηρεσία και γι' αυτό γίνεται μια δεύτερη αποστολή. Ε, φαίνεται ότι υπήρξε μια οργανωμένη εκστρατεία κατά της ε, ε, υπηρεσίας αυτής, αλλά δεν ήταν όλοι οργανωμένοι οι γονείς που θέλανε να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των παιδιών τους. Ε, δεν λένε ότι όλοι είναι ανήκαν σε αυτήν την υπηρεσία ή όλα όσα κάνει η υπηρεσία είναι λάθος. Δεν μπορούμε να λέμε επίσης με τον ίδιο τρόπο ότι όσοι έχουν υπογράψει την αναφορά κάνουν μια εκστρατεία κατά της υπηρεσίας. Σε αυτούς τους έξι μήνες λοιπόν προσπαθήσαμε να βρούμε μια συμβαστική λύση ως προς τη σύνταξη συστάσεων στις γερμανικές αρχές και δεν έχουμε καταφέρει να να φτάσουμε σε κοινό συμπέρασμα. Έχουμε ανταλλάξει τόνου ε, email και γνωμοδοτήσεων, έχουμε συζητήσει, αλλά ποτέ δεν φτάσαμε σε συνένεση. Η Επιτροπή Αναφορών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η οντότητα που είναι όσο πιο κοντά γίνεται στους Ευρωπαίους πολίτες σε σχέση με τις υπόλοιπες. Έχουμε ανθρώπους ε, που έρχονται σε εμά από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για διάφορα θέματα. Όταν γίνεται παραβίαση ενός άρθρου της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, ειδικότερα σε ευαίσθητα θέματα σαν αυτό, ε, οι άνθρωποι επενδύουν σε μας τις προσδοκίες τους. Είμαστε, ας πούμε, η τελευταία, το τελευταίο καταφύγιο για αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό αποφασίσαμε ότι πρέπει να αλλάξει η διαδικασία ε, σε αυτό το ε, ιδιαίτερα συζητημένο και δύσκολο θέμα. Δεν μιλάω εκ μέρους όλων, ειδικότερα όσων δεν είναι εδώ σήμερα, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε δύο κείμενα. Το ένα είναι η δική μου έκθεση, αυτή που έγραψα εγώ. Και να πω ότι έχω συμπεριλάβει σχεδόν όλες τις απόψεις των ε, ε, συναδέλφων και η δεύτερη είναι αυτή της γραμματείας. Ε, ποια θα είναι η μοίρα αυτών των κειμένων στο εξή. Εμείς θα το αποφασίσουμε. Ε, είναι ιδιαίτερα πιστικό παρόλα αυτά το γεγονός ότι εάν καταθέσουμε προτάσεις τροπολογιών για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα όπως αυτό, αν αυτό γίνεται από ανθρώπους που είτε δεν είναι εδώ σήμερα ή δεν πήγαν ποτέ στις αποστολές στο Βερολίνο ή δεν εκεί έμαθαν τις πληροφορίες που μας έδωσαν οι γερμανικές αρχές, ε, δεν ξέρω. Ε, οι πληροφορίες ε, που δόθηκαν στο Περολίνο ήταν κάπως ελλειπής θα έλεγα. Δεν μπορέσαμε να φτάσουμε σε κάποια ουσιαστικά συμπεράσματα για το αν υπήρξε παραβίαση ή όχι. Αλλά αυτός δεν ήταν ο σκοπός μας. Ε, ο σκοπός μας ήταν να βρούμε γεγονότα και να βοηθήσουμε τους πολίτες αυτούς. Μέχρι το, από το τέλος της ε, αποστολής και μέχρι σήμερα συνεχίζουμε να λαμβάνουμε email, τηλεφωνήματα, επιστολές και αναφορές από ανθρώπους που ε, έχουν πληγεί από τη δράση της Jugendamt. Έτσι λοιπόν είτε επιλέγουμε την ε, γραμματεία που επιτρέπει ε, το κείμενο της γραμματείας που επιτρέπει τροπολογίες ή επιλέγουμε το δικό μου κείμενο ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας και πάλι θα αποφασίσουμε για μια καταλεκτική ημερομηνία για το τελικό κομμάτι του κειμένου ως προς την κατάθεση τροπολογιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την ε, η συγγήτρια, Από την πλευρά της γραμματείας να πω ότι χθε ε, ενημερώθηκαν οι βουλευτές με email ότι σήμερα θα γίνει η συζήτηση το απόγευμα και όχι το πρωί. Έτσι λοιπόν η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι Παρασκευή 11 Μαΐου. Η έκθεση θα ψηφιστεί στην ε, συνεδρίαση μας τον Ιούνιο. Τώρα λοιπόν να σας πω ότι η λίστα των ε, αναφορών Β πρέπει να περάσει στην Α. Το, σημείο 19, 23, 22 και 21 και έτσι κλείνει η συνεδρίαση. Κυρία Γιωτοβά, έχετε για άλλη μια φορά το λόγο. Νομίζω ότι πρέπει να ψηφίσουμε για το κείμενο που θα επιλέξουμε. Το κείμενο της γραμματείας ή το κείμενο που συνέταξα εγώ. Η γραμματεία ότι δεν θα, ε, ε, λέει ότι δεν θα ασχοληθεί με το θέμα. said the amendment should be to the Secretariat so that they can add to it. And they have received the Secretariat. And they've received it. You should say, Mr. Just take the floor. It was the understanding that the από άποψη διαδικασίας η λύση θα ήταν να ψηφίσουμε το κείμενο της γραμματείας που είναι ο κοινός παρανομαστής μεταξύ όλων των μελών της Επιτροπής ε, ως τώρα, αλλά αναγνωρίζει ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποια επιπλέον σημεία που θέλουν κάποια μέλη να προσθέσουν και αυτά θα πρέπει να τα ε, προσθέσουμε ως τροπολογίες. και να μην ασχοληθούμε με ένα κείμενο που, δεν έχει ένα κοινό που να μην είναι κοινό παρανομαστής. Νομίζω ότι λοιπόν αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσαμε το μεσημέρι της Παρασκευής είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες και τα επιπλέον σχόλια στο κείμενο αυτό. Παρακαλώ για σχόλια. κυρία Σκολάρσκαβης. Συναντήσαμε τα μέλη της αντιπροσωπείας στο Στρασβούργο. Όλοι μας, οι οποίοι ήμασταν παρόντες, το συζητήσαμε αυτό το θέμα και ψηφίσαμε για ποιο κείμενο θα ήταν το σημαντικό και αποφασίσαμε ότι κύριε Γιωτόβακεκ. Λοιπόν, δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει, διότι μέχρι τώρα πίστευα ότι δουλεύαμε πάνω σε αυτό το κείμενο και εγώ ετοιμάζω τροπολογίες για αυτό το κείμενο. Και τώρα εντωμεταξύ κάτι έχει αλλάξει. Μπορείτε να μου πείτε τι άλλαξε τελικά, εντωμεταξύ. Domnule ε, Macmillan Scott, aveți cuvântul. Ζητώ συγγνώμη που δεν ήρθα νωρίτερα, ειλικρινά. Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ λεπτό και ευαίσθητο και στο συγγνώμη. Επειδή ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια και αντιλαμβάνομαι πλήρως τα διάφορα συμφέροντα που εκπροσωπούνται εδώ σε αυτή τη γνωμοδότηση. Νομίζω όμως για μένα τουλάχιστον το πρόβλημα είναι δεδομένου ότι λάβαμε αυτά τα κείμενα τώρα και τώρα ζητείτε να ε, κατατεθούν τροπολογίες για την Παρασκευή, έχω την εντύπωση ότι η ομάδα θα προτιμούσε να έχει λίγο περισσότερο χρόνο. Δεν ξέρω πόσο επίγον είναι το θέμα, διότι για ένα τόσο σημαντικό θέμα και με βάση τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της ε, Συνθήκης της Λισαβόνας που εισάγει για πρώτη φορά ε, νέες έννοιες για τα δικαιώματα των παιδιών, Πρόεδρε, αναρωτιέμαι κατά πόσον μπορείτε να μας δώσετε λίγο περισσότερο χρόνο, ώστε οι ομάδες και το Κοινοβούλιο να εξετάσουν αυτό το ευαίσθητο και σημαντικό θέμα. Δεν ξέρω πόσο επίγουν το θέμα, εσείς θα μου πείτε. Ο κύριος Μποστινάρο. Ευχαριστώ. Σήμερα το πρωί είχαμε συζητήσει για το θέμα της ενημέρωσης στη Ρουμανία. Πρέπει να καταλήξουμε σε μία συνένεση. Είχαμε βρεθεί αρκετά κοντά σε μια συμφωνία και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Δεύτερον, όποια και αν είναι η έκθεση που θα γίνει δεχτή, δεν θα πρέπει να είναι αντίθετη ε, προς τον βασικό προσανατολισμό της έκθεσης που έχει συντάξει ο εισηγητής διότι η πρόεδρος της αντιπροσωπείας ήταν η κυρία Ματσόνη. Εκείνη λοιπόν είναι εκείνη που πρέπει να μας πει ποια θα είναι η δομή της έκθεσης και εμείς μετά θα αντιδράσουμε ανάλογα με αυτά που θα μας πει. Δεν πρέπει από τη γραμματεία να έρχεται κάτι το οποίο θα είναι αντίθετο με αυτά που πιστεύει ο εισηγητής. Ελπίζω να κάνουμε αυτό που έγινε και σήμερα το πρωί, δηλαδή να ακολουθήσουμε το προσανατολισμό ε, της κυρίας και να συντάξουμε μια έκθεση της ενημερωτικής επίσκεψης της Επιτροπής και όχι ε, διάφορες εκθέσεις ηγετών κατά της αντιπροσωπείας και το αντίστροφο, διότι αυτό θα δημιουργήσει περιττές εντάσεις και διαφορές. Παρακαλώ λοιπόν ειλικρινά, επιμένω, να συνεχίσετε να εργάζεστε Φροντίζοντα χρειάζεται, φροντίζοντας ο προσανατολισμός να είναι πάντοτε εκείνος που προτείνει ο εισηγητής. Μετά, οι αποχρώσεις, λεπτομέρειες δεν έχουν σημασία. Αλλά τελικά θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλει ο εισηγητής. Λοιπόν, μετά από τα όσα άκουσα θα πρέπει να τα δούμε με τα μέλη και τη γραμματεία και θα επανέλθουμε σε εσά με λεπτομέρειες για την διαδικασία που θα υιοθετηθεί. Έχετε το λόγο. Να συμπληρώσω κάτι ως τώρα. Αναγνωρίζω ότι η έκταση για την οποία μιλάμε, αυτή της γραμματείας, δεν ε, είναι αντίθετη σε καμία περίπτωση. Εγώ προσωπικά θα προτιμούσα αν πολύ γρήγορα και με συνοπτικό τρόπο, με πιο συνοπτική μορφή, είχαμε τον πυρήνα. Δεν είναι λοιπόν ε, κάτι αντίθετο, είναι μία έκδοση που είναι χρήσιμη στην όλη διαδικασία. Αυτή είναι η δική μου αξιολόγηση που ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι η μία, μία έκδοση που είναι κατά της άλλης έκδοσης, η κυρία Γιώτοβα. Αγαπητοί συνάδελφοι, κατανοώ πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το θέμα. Έχουμε ε, διαφιλονικές ακόμα και εδώ στην Επιτροπή. Πολλοί από αυτούς που είναι παρόντες εδώ δεν γνωρίζουν ακριβώς ε, σε τι αναφερόμαστε. Η έκθεση που έχω καταθέσει δεν έχει ως στόχο να επιλύσει αυτό το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα. Πρόκειται για μια έκθεση η οποία βασίζεται στα όσα είδαμε, ακούσαμε και να αναλύσαμε κατά τη διάρκεια της αποστολής. Και λάβαμε υπόψη τις προτάσεις, τις τροπολογίες που πρότειναν οι συνάδελφοι, τα μέλη της Επιτροπής. Θα ήθελα να σας ζητήσω, όποια συζήτηση και αν γίνει για τα δύο κύματα, όπως είπε η κυρία Μποβισκά, θα πρέπει να έχουμε και την γνώμη των, της αντιπροσωπείας. Συναντηθήκαμε με αυτούς και με ψηφοφορία αποφασίσαμε στο Στρασβουργό πώς θα εργαστούμε και όλοι έδειξαν ότι προτιμούν τη δική μου έκθεση. Κυρία Μποβίνσκα, τελευταία λόγια. Είπατε ότι θα διαβολευτείτε με τη γραμματεία, τα άλλη μέλη κτλ. Χρειαζόμαστε έναν πιο διαφανή τρόπο διαβούλευσης. Το θα διαβολευτούμε με τον ένα και τον άλλον δεν ξέρω με ποια μέλη, με ποια διαδικασία και πώς θα ληφθεί η απόφαση. Θα ήθελα κάπως, τέλος πάντων, να ενημερωθούμε για το πώς θα ληφθεί αυτή η απόφαση, γιατί εγώ θεωρούσα ότι είχε ληφθεί η απόφαση και τώρα βλέπω την άλλη απόφαση. Θέλω απλώς να μάθω ποιες είναι οι διαδικασίες. Uh, Μετά από αυτή την ε, συζήτηση θα πρέπει μάλλον να οργανώσουμε άλλη μία συνάντηση για να μπορέσουμε να συζητήσουμε αυτή την έκθεση. Άρα εσείς ε, θα πρέπει να ε, θεσπίσετε το νέο ραντεβού. Κλείνει η συνεδρίαση.